Ο προσκεκλημένος από την Αυστρία βρίσκεται εδώ. Κοιτάξτε να ξεκινήσουμε με τη τα διάταξη διότι είναι πολύ φορτωμένο. Σας καλωσορίζω και θα ήθελα να προτείνω κάποιες αλλαγές στη μέσα μετά από αιτήματα των εμπλεκομένων συναδέλφων. Πρώτα απ' όλα να σας ζητήσω να συμφωνήσετε πως το σημείο υπάρχει μόνο 7 γνωμοδότηση του Βλάσακ για την ελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας να εξεταστεί πριν από το σημείο 5 της Μεσσίας Διατάξεως. Ως εκ τούτου θα διεξαχθεί η συζήτηση 4 η ώρα και το θέμα που αφορά στην ενιαία αγορά για τις επιχείρησεις για την ανάπτυξη στο σημείο 5 θα εξεταστεί μετά από το σημείο 7. Το για αύριο να σας πω ότι η ώρα ψηφοφοριών θα καθυστερήσει κατά 30 λεπτά Δηλαδή θα ξεκινήσουν, μάλλον θα ε, διεξαχθεί στις 30, δηλαδή θα προταχθεί κατά 30 λεπτών. Λοιπόν, και το σημείο που αφορά στην Ρουμανία θα εξεταστεί ως τελευταίο σημείο της μισής τετάξης. Τώρα, αν δεχόσετε τις αλλαγές, γιατί δεν υπάρχουν άλλες αιτήσει για τροποποίηση, να πούμε ότι εγκρίνει τη μισή διάταξη. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 2 τη μισή η έγκριση των πρακτικών τη 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2010 και τη 9η Δεκεμβρίου. Τα πρακτικά ω συνήθω έχουν διανεμηθεί, είναι διαθέσιμα και θα θεωρήσουμε πως ε, έχουν εγκριθεί το τέλος της συναδριάσεω. Περνάμε στο σημείο 3 τη Συμβουλευτικής Διατάξεω, αν φυσικά δεν έχουν πάρει τι ενστάσει. Ε, περνάμε στο σημείο 3 λοιπόν που είναι η ανακοινώση τη Προέδρου. Να σα πω ότι σήμερα έχουμε ανάμεσά μας μια ομάδα επισκεπτών. Είναι ιδιαίτερη σημασία ε, επισκέπτες. Του προσκαλέσει ο συνάδελφος Κέλλη. Είναι φοιτητέ ε, από το Κόρκ και τους υποδεχόμαστε με ένα χειροκρότημα. Να πω και κάτι ακόμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εργασίες της Επιτροπής μας αλλά και για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Να σας ενημερώσω ειδικά όσους δεν είναι μέλη της Επιτροπής ΣΟΥΡ ότι στις 10 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 στην Επιτροπή ΣΥΟΡ προγραμματίζεται μια συνεδρίαση για την πολιτική συνοχή. Στην Επιτροπή λοιπόν θα εξετάσουμε όλα τα σημαντικά θέματα που άπτονται της πολιτικής συνοχής. Θα υπά... συμμετάσχει και ο Επίτροπος Χάν, θα υπάρχουν πολλοί ε, ομιλητές, συντονιστές, αλλά και πολύ και όσοι εξημών μάλλον θέλουν να συμμετάσχουν στην συζήτηση, να προετοιμαστείτε καταλήλως και να χρησιμοποιήσετε ως βάση τα έγγραφα που έχουμε γκρίνει ως Επιτροπή Ρέτζο. Θα είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική συνάντηση. Η συζήτηση επίση θα έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι θα μπορέσει να επηρεάσει και τις απόψεις ε, της Επιτροπής του ΣΟΥΡ. Τώρα να περάσουμε το σημείο 4 της μισής Διατάξεως. Ε, πρόκειται για την έκθεση του κυρίου Μίλιοσλαβ Μικολάσικ ε, σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων πολιτικής για το έτη 2007-2013. Ο Μύροσλαβ έχει προσκαλέσει για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και κάποιον ο οποίος έχει εμπλακεί εδώ και πολλά χρόνια επικοδομητικά στην διαμόρφωση της ε, πολιτικής συνοχής, τον Ζάνης Ροσμπάχερ, υπεύθυνο για την, ε, την της Αυστρίας ε, για την διάσκεψη χωροταξικού σχεδιασμού στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω την έκθεση. Το κείμενο ελπίζω να γίνει δεκτό. Ήρθα σε επαφή με όλους τους συζητητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και συμφώνησαν με τις αρχικές μου σκέψεις. Θα ήθελα να σας ε, αναφέρω τι έχω προετοιμάσει για τη σημερινή συνεδρίαση και όπως είπε η κυρία Πρόεδρος Ντανούτα Χιούμπνερ θα έχουμε και έναν ε, εμπειρογνώμων από την Αυστρία άρα θα ακούσουμε μια σειρά από θέσεις ε, σήμερα η ανακοίνωση τη Κομισιόν με τίτλο Πολιτική Συνοχή στα ειδική έκθεση 2010 σχετικά με την εφαρμογή του πρόγραμμα των 2007-2013 ως έγγραφο εργασία του εσωτερικού της Κομισιόν αναφέρεται στα αποτελέσματα από την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Αυτή είναι και η πρώτη ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να αναλύσει και να αξιολογήσει τη διαδικασία υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που ξεκίνησαν το 2007. Ταυτόχρονα αποτελεί και την ευκαιρία προκειμένου το Κοινοβούλιο να εκφραστεί επί του Πώ πόσο τα κάρτε δεσμεύτηκαν στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος και στις δαπάνες. Εάν ε, θεωρούμε ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εφήρμοσε ε, τα προγράμματα αυτά. Η έκθεση λοιπόν αυτή αφορά στην εφαρμογή των προγραμμάτων ε, κατά την προγραμματική περίοδο και στην στρατηγική ε, ενημέρωσης και πληροφόρησης που αφορά επίσης στο μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής. Εφαρμογή των προγραμμάτων. Συντομία. Το, ο το, τα κονδύλια ανέρχονταν σε 93,4 δις ευρώ για την περίοδο, κάτι που του επιτελεί πάνω από 24, 27% των διαθέσιμων πόρων για την περίοδο. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τα κράτη-μέλη ε, μπορεί να θεωρηθεί εύλογη λαμβάνοντας υπόψη ε, της, ε, την επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης τα έτη 2008-2009 οφειλόμενη στην ε, παγκόσμια κρίση αλλά και στις μεταρρυθμίσεις ε, που έγιναν την περίοδο 2007-2013. Πάντως κάποια κράτη-μέλη ε, είναι κάτω από το 27% που είναι ο Ευρωπαϊκό μέσος όρος και οι διαφορές είναι σημαντικές ανάμεσα στα κράτη και ανάμεσα στις, στα διάφορα, στις διάφορες θεματικές πολιτικές. Έχουμε ε, ποσοστά κάτω του 20% για τέσσερα κράτη-μέλη. Ε, αυτό το, αυτός ο μέσος όρος ε, έχει, διαφοροποιείται ανάλογα με τους στόχους σύγκληση, αγωνιστικότητα, απασχόληση και εσωτερική συνεργασία. Επίσης εφαρμόζεται και στο ποσοστό των κονδυλίων που έχουν δοθεί για τις που έχουν κρατηθεί μάλλον ε, στις διάφορες πολιτικές. Αφού μελετήσαμε τα σχετικά στοιχεία, θεωρώ ότι περισσότερο προσπάθειες χρειάζεται να καταβληθούν σε ορισμένους τομείς, ειδικά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της, ε, και βελτίωση της εφαρμογής, να αποφύγουμε ε, υπερβολικές καθυστερήσεις, να και τέλος να αυξήσουμε τις συνέργειες ε, με άλλες ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να επιταχυνθούν λοιπόν η εφαρμογή και η υλοποίηση του προγράμματος ιδιαίτερα στον τομέα των ε, σιδοδρόμων, στις επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, στην θέμα της ικανότητας δημιουργίας, δυνατότητας δημιουργίας ικανοτήτων κλπ. Επίσης, η εφαρμογή των προγραμμάτων είναι μια διαδικασία συνεχής και δυναμική, η οποία μπορεί να επηρεαστεί από τον εντοπισμό κάποιων ελλείψεων ε, στους διάφορους κλάδους ε, όπου απαιτούνται μεταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστούν οι βέλτιστες πρακτικές, κάτι το οποίο δεν να, βοηθήσει μάλλον τους άλλους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα. έκθεση λοιπόν ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να διορθώσουν τις καθυστερήσεις σε ρηφορά την επένδυση των πόρων και να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικά προγράμματα για να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 2. Τι αναφορέ σχετικά με τη στρατηγική. Αυτό είναι ένα εργαλείο για την συζήτηση των θεματικών διαστάσεων, των πολιτικών που βασίζονται σε ε, στοιχεία τα οποία υποβάλλουν τα κράτη-μέλη. Η στρατηγική αξιολόγηση αποτελεί και μια διαδικασία αξιολόγησης των, ε, της όλης ε, διαδικασίας προκειμένου να έχουμε μια γενική άποψη της κατάστασης και ε, έχουμε τις απαραίτητες βάσεις για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την απόδοση. Θα όμως να τονίσω κάποιες καλές, κάποιες χρηστές πρακτικές οι οποίες συμβάλλουν στην ε, βελτίωση της, ε, του όλου εγχειρήματο και βελτιώνουν την θέση των εμπλεκομένων στα κρατημέλη. Καλύτερε στρατηγικέ είναι οι εξή. Χρησιμοποιούνται κάποιοι δείκτες ε, κεντρικοί να είναι αναφορά και ενημέρωση σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ εθνικών πολιτικών και κοινωνικών πολιτικών, οργάνωση δημοσίων συναντήσεων και συζητήσεων με τους εμπλεκομένους υποβολή ε, νομοδοτήσεων και εκθέσεων προς τα Εθνικά Κοινοβούλια και η δημοσίευσή του στο διαδίκτυο. Όπως ε, βλέπετε προσπαθώ να είμαι το δυνατόν σύντομος διότι ελπίζω πως θα ακολουθήσει μια ε, ικανοποιητική συζήτηση. Φτάνω λοιπόν στα συμπεράσματα προτού να, λάβουν το λόγο, να λάβει το λόγο ο ειδικό προσκεκλημένος έκθεση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την ε, βελτίωση της πολιτικής συνοχής ε, αυτήν την ενδιάμεση περίοδο. Επίσης ε, χρειάζεται να φροντίσουμε να βελτιώσουμε τις επιπτώσεις της κοινωνικής συνεχής και να συμβάλλουμε στην ε, ολοκλήρωση αυτής της πολιτικής. Καταλήγω να πω ότι πιστεύω πως η μελλοντική μας συνεργασία θα συνεχίσει να είναι επικοδομητική και θα συμβάλλει στην ε, ε, υψηλή αποτελεσματικότητα και ποιότητα της πολιτικής της έκθεσης που θα ολοκληρωθεί το 2013. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω τον πισεκλημένο ομιλητή. Πρόκειται για τον κύριο Ιωχάνης Ροσμπάχερ, βρίσκεται στα δεξιά μου. Ευχαριστώ κύριο Ροσμπάχερ. Ο κύριος Ροσμπάχερ θα μας μιλήσει για το θέμα και θα μας μιλήσει για την εμπειρία του στον, ε, στη θέση που καλύπτει τώρα. Παρελθόν είχε δουλέψει στην ε, Βρυξέλλες και προηγούμενα ήταν και ομοσπονδιακό ήταν εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας ε, στις Βρυξέλλες και τώρα συμμετέχει στην Αυστριακή Διάσκεψη Χορταξιδισμού της οποίας και είναι διευθυντής. Ε, ευχαριστώ κύριε Ροσμπάχερ, έχετε το λόγο και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς υπάρχουν ε, μικροφωνισμοί. Υπάρχει πρόβλημα με τα μικρόφωνα. Κάποιος θα έπρεπε να κλείσει το μικρόφωνο του παρακαλώ. Please, I hope so. So, noch einmal, ja, jetzt ging es besser. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα και τους συναδέλφους από το Συμβούλιο που είναι παρόντες. Όταν ο κύριος Μικολάσικ με παρουσίασε. Ήταν τότε εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Βλέπω λοιπόν πολλούς ανθρώπους, την κυρία Κρέλ, τον κύριο Όλμπρεχ, τον κύριο Φωνής Λερόι, που τους είχα γνωρίσει στο παρελθόν, κάποιους σε άλλες, ε, υπό άλλες ιδιότητες. Εν πάση ο στόχος μας δεν είναι να μιλήσουμε για το παρελθόν, με καλέσατε. Ελπίζω να πω κάτι για αυτά τα οποία αφορούν την στρατηγική προσέγγιση για τα περιφερειακά θέματα και τι μπορούμε να προσθέσουμε, τι μπορούμε να συνεισφέρουμε στα κράτη-μέλη με αυτήν την ε, λογική. Θα κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις μετά τρία slides τα οποία έχουν να κάνουν με τη στρατηγική σύνταξη εκθέσεων στην Αυστρία ιδιαίτερα μια ειδική εφαρμογή το strat στην Αυστρία και επίση θα δούμε τι προβλέπεται για το μέλλον επέκεινα του 2014. Ε, εγώ δεν ξέρω πολύ καλά τα άλλα κράτη-μέλη, ξέρω, ελπίζω ότι η δική μου χώρα, η, η Αυστρία είναι μια χώρα η οποία έχει 8,4 εκατομμύρια ε, κατοίκων ε, περίπου πυκνότητα 100 κάτι για ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, αλλά αυτό δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονό ότι ένα μεγάλο μέρο τη Αυστρία είναι βουνά και δεν είναι κατοικήσιμο. Έχουμε 9 περιοχέ στην Αυστρία και έχουμε 8 γειτονικέ χώρε. Και αυτό φυσικά έχει κάποιε επιπτώσει στην χρήση των ε, περιφερειακών πόρων. Ο στόχος της πολιτικής μας είναι να έχουμε ε, μία γενική υποστήριξη βάσει των διαρθρωτικών στόχων, στο ανατολικό μέρος έχουμε και μια περιοχή η οποία εμπλέκεται στους στόχους σύγκλησης. Έχουμε το Strategic Reference Framework, την Εθνική Στρατηγική, που περιλαμβάνει 21 λειτουργικά προγράμματα. Η συνολική χρηματοδότηση είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σχεδόν, που είναι περίπου 0,4% του συνολικού ταμείου συνοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε δεν είναι πολλά χρήματα. Γιατί έχουμε 21 λειτουργικά προγράμματα, έχουμε όπως σα είπα 9 περιφέρειες, έχουμε δύο προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου και στη συνέχεια 10 προγράμματα εδαφικής συνεργασία για να, συνεργαστούμε με τους γειτονές μας, μεταξύ των οποίων τρία είναι ε, διαμεθοριακά είναι προγράμματα που εμπλέκουν παραπάνω από ένα κράτος, είναι περιφερειακού χαρακτήρα. Επίσης, για να δείτε τι μπορούν να επιτύχουν οι περιφερειακοί πόροι, τα 200 εκατομμύρια που παίρνουν κάθε χρόνο είναι 0,08 του ΑΕΠ της χώρας μας, της Αυστρίας. Περίπου 0, αν θέλετε. Μια δεύτερη επεξήγηση που θέλω να κάνω. Τι καινούριο μας έχει φέρει αυτή η χρονική περίοδος η οποία είναι το αντικείμενο αυτής της ε, παρουσίασης. Έχουμε τρία στοιχεία. Η συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εθνικές στρατηγικές στα κράτη-μέλη. Για μας είναι γνωστό αυτό ως στρατ η Εθνική Στρατηγική και υπάρχει και η δημιουργία εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο 2009 και 2012 σε εθνικό επίπεδο και επίσης για προγράμματα υπάρχουν αιτήσει εκθέσεις, εκθέσεις λογιστικού απολογισμού κτλ. Εγώ θεωρώ και τολμώ να πω ότι τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση έχει επιτύχει αυτή η διαδικασία για τις στρατηγικές εκθέσεις. Έχουμε λοιπόν συντάξει μια έκθεση όπως και τα άλλα κρατημέλη. Έχω φέρει μερικά, έντυπα, μερικά αντίτυπα μαζί σας εάν θέλετε, αλλά μπορείτε να το πάρετε και σε ηλεκτρονική μορφή στα αγγλικά. Έχουμε δημοσίευση λοιπόν αυτή την έκθεση. Και ποια είναι τα κύρια πορίσματα τώρα αυτής της έκθεσης. 22% ε, απορρόφηση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009. Σας φαίνεται λίγο λίγο αυτό. Και έχετε δίκιο άμα το δείτε έτσι απομονωμένα. Αλλά παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε απορροφήσει όλα τα χρήματα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πολύπλοκα προγράμματα τα οποία χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε θεσπίσει ένα πολύ καλό πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσει. Όπως βλέπετε, έχει σχεδόν διπλασιαστεί η απορρόφηση, μάλλον έχει πάνω από διπλασιαστεί η απορρόφηση μέχρι την πρώτη του 2011 που έχει φτάσει σε 48% η απορρόφηση. Ένα άλλο στοιχείο είναι αντίθετα με την ε, γενική σχεδίαση έχουμε μια ιδιαίτερη εστίαση στις επιχειρήσεις αυτό οφείλεται και στην οικονομική κρίση υπήρξε ανάγκη να ενισχυθεί ο επιχειρηματικό σύστος και αυτό φυσικά είχε και κάποιες επιπτώσει στο ύψος της ε, απορρόφησης. Τα προγράμματα τα οποία ήταν ε, καινοτόμα ε, είχαν ιδιαίτερο ρόλο. Η Αυστρία βέβαια είναι μια πλούσια χώρα όταν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, αυτό ήδη θα έχει αντιμετωπίσει και αντικείμενο εθνικής ε, πρόνοιας. Οι διαφορετικοί πόροι προσθέτουν ακόμα ένα όροφο στο οικοδόμημα της κρατικής ε, ε, λειτουργίας στα θέματα αυτά. Και τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια έγιναν θετικά αποδεκτά λόγω και της κρίσης. Ένα τέταρτο σημείο υπήρξε με αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια έκθεση σε σχέση με τις περιοχές που πλήττονται από την οικονομική κρίση και τι έχει κάνει το πακέτο αυτό των διαρθωτικών πόρων για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Και το αποτέλεσμα της ε, έρευνάς μας ήταν ότι λειτουργήσαν καλά αυτά τα προγράμματα και δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική αλλαγή στρατηγική που ακολουθήθηκε, απλώς μονάχα μικρές προσαρμογές στα προγράμματα. Τώρα, έχουμε μια σειρά από προκλήσεις που ακόμα πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στην προσπάθειά μας και φυσικά θα πρέπει να επιζητήσουμε και μεγαλύτερη ορατότητα. Αυτό είναι δύσκολο όταν δεν έχουμε αρκετά χρήματα, αλλά είναι στόχοι που θέλουμε να του επιτύχουμε. Μας ενδιαφέρει επίσης σε τομείς οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην πολιτική συνοχής Μιλάμε για έρευνα και ανάπτυξη, μιλάμε για ε, εκκίνηση επιχειρήσεων και ο στόχος μας είναι μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των τομέων. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το θέμα της απλοποίησης και αυτό βρίσκεται υπό <clears throat> τροποποίηση στους αντίστοιχους, πολλά βρίσκονται υπό απλοποίηση στους κανονισμούς ο στόχος μας ήταν να έχουμε απλοποίηση της δομής του κόστους με ποσά κατά τα λοιπά. Θέλησαμε να τα εφαρμόσουμε αυτά περισσότερο στην Αυστρία και να περιληφθούν στα προγράμματα αυτά. Αυτό πήγε και αυτό καλά. Τα διδάγματα τα οποία έχουμε αποκομίσει τώρα. Εμείς μπορούμε να το δούμε αυτό το θέμα μόνο από την οπτική γωνία της Αυστρίας. Και η εντύπωση μας είναι ότι ακόμα και αν ήμασταν κάπως σκεπτικιστές σε σχέση με αυτό το πρόσθετο επίπεδο στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, η παρουσία των ε, κοινοτικών προγραμμάτων μας έχει βοηθήσει. Έχουμε, όπως ξέρετε, 21 προγράμματα και με πολλά από αυτά έχουν διευρυνθεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι σημαντικό γιατί είναι η πρώτη φορά που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια γενική γραμμή και έπρεπε κάπως να κατευθύνουμε τους πόρους αυτούς της πολιτικής συνοχής με βάση τους στόχους της Λισαβόνας, δηλαδή ο λεγόμενος προσδιορισμός της Λισαβόνας. Μας ενδιαφέρει επίσης να εξασφαλίσουμε τη συγκρισιμότητα, να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, να καθορίσουμε καλύτερα τους χώρους παρέμβασης, γιατί τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να πάρουν μια απόφαση για το πού θα επενδύσουν και επομένως θα ήταν απαραίτητο να υπάρχει μια σειρά δικτών που θα μας βοηθούσαν να έχουμε μια καλύτερη κατεύθυνση και που θα μας θα επέτρεπαν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια καλύτερη εικόνα για την, ε, τις κατευθύνσεις των ε, χρηματοδοτήσεων. Βέβαια, υπάρχουν όρια, οι εκθέσεις αυτές δεν είναι ο ντέος εξμάκινα, δεν είναι πανάκια που λύνει όλα τα προβλήματα. Όταν, παραδείγματο χάρη, λέει η Κομισιόν ότι δεν υπάρχει τροποποίηση των ε, περιφερειακών ανισομεριών, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ δύσκολο να καταμετρηθούν όλα αυτά και να αντιμετωπιστούν. Έχουμε πάρα πολλά αριθμητικά στοιχεία, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε επιπλέον και πρέπει να καταλήξουμε σε μια καλή ισορροπία μεταξύ της παρουσίασης επί τη βάση των ε, δικτών και της ε, ποιοτική ε, περιγραφής και αξιολόγησης για το μέλλον. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. μιλάω για την αυστριακή προσέγγιση και είμαστε πολύ περήφανοι για όλα αυτά. Όπως σας είπα, είμαστε <clears throat> υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε αυτή τη στρατηγική. Υπήρξαν όλες αυτές οι εκθέσεις οι οποίες σας ανέφερα ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε και μια συνοδευτική διαδικασία εποπτείας για τα θέματα αυτά. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με υποχρεωτική βάση, γίνεται εθελοντικά και εδώ έχω αναφέρει ορισμένα σημεία που περιγράφονται και στην ε, έκθεσή μας εδώ πέρα, αν θέλετε να τη διαβάσετε. Ο στόχος είναι η κοινοτική πολιτική, η πολιτική λοιπόν αυτή και η τοπική εμπειρογνωμοσύνη να μπορέσουν να έρθουν από κοινού περισσότερο, να υπάρχει μια μεταλαμπάδευση πληροφοριών, να συνδεθούν με το πολιτικό επίπεδο και να υπάρξει μια μεγαλύτερη, ένας μεγαλύτερος διάλογος και να αναπτυχθούν στρατηγικές, ε, στρατηγικού χαρακτήρα συζητήσεις. Έχουμε χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες δομές, δεν δημιουργήσαμε περαιτέρω φορείς. και χρησιμοποίησαμε τις ε, δυνατότητες που είχαμε σε οικονομικό επίπεδο για να διοργανώσουμε συνέδρια όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και αυτό έτυχε μια πολύ καλή αντιμετώπιση. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το μέλλον. Όπως είπαμε, από την αυστριακή πλευρά θεωρούμε ότι το εγχείρημα αυτό είχε ένα σημαντικό ενδιάμεσο χαρακτήρα γιατί μπόρεσε να υπάρξει μια παρέμβαση μεταξύ όχι μόνο του ευρωπαϊκού και του περιφερειακού επίπεδου αλλά και μεταξύ διαφορετικών οικονομικών τομέων μπορέσε να δουλέψει ως συγκολητικό συστός επομένως το εγχείρημα αυτό Η Κομισιόν αναφέρεται στον ΤΥΠΚΟ στην εταιρική σχέση για την συνεργασία και την ανάπτυξη. Πιστεύω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούν τα οι προσπάθειες αυτές και για το δεύτερο σημείο, για την ε, σύνταξη εκθέσεων, είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Για να υπάρχει μια σωστή έκθεση, η έκθεση αυτή απαιτεί χρόνο. Και αυτό αφορά όλες τις εκθέσεις, είτε είναι λογιστικοί απολογισμοί ή κάτι άλλο. Και αυτό αφορά, φανταζόμαι, και τις ε, προτάσεις της Κομισιόν για τις ε, χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις, όπου πολλές φορές η Κομισιόν είχε εξωπραγματικές απαιτήσει. Πάρα πολλά από αυτά εμπλέκονται στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 ή θα έχουμε εκθέσεις οι οποίες είναι αυστηρά εναρμονισμένες στον χρόνο ή θα έχουμε εκθέσεις οι οποίες είναι καλές σε επίπεδο περιεχομένου και αυτό αφορά όλε τις εκθέσεις. Μια στρατηγική έκθεση ετησίου χαρακτήρα στην πράξη απαιτεί μισό χρόνο. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε λοιπόν για όλα αυτά. Εμεί θα θέλαμε περισσότερο να μιλήσουμε για συντονισμό των διαφόρων φορέων και ε, ενεργειών και όχι για συντονισμό, γιατί ο συντονισμός δίνει την εντύπωση ότι κάποιος εκ των άνω προσπαθεί να επιβάλλει ένα τρόπο λειτουργίας. Ο χρόνος λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, για την ε, αποτελεσματόστροφη αντιμετώπιση δεν έχω να πω κάτι άλλο και για το... Σας είπα ότι υπάρχει το τελικό αποτέλεσμα και το outcome και το <laughs> αποτέλεσμα. Η χώρα μου έχει μια πλούσια γλώσσα, αλλά δεν έχουμε κάτι στα γερμανικά για τη λέξη outcome. Δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να το πω στη γλώσσα αυτή και όταν δεν ξέρουμε τι ακριβώς βρίσκεται πίσω από μια λέξη, μια τέτοια λέξη δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι η πιο πρόσφορη διατύπωση για την πολιτική από το 2014 και επέκεινα. Η πολιτική αυτή δεν μπορεί να είναι ένας μοχλός που τον τραβάμε και δουλεύει το μηχάνημα. Είναι σαν ένα τεράστιο πλοίο το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δουλεύει μαζί για να το κάνει να κινηθεί. Όταν πρέπει να έχουμε μια μεθοδολογία την οποία θέλουμε να καταλαβαίνουμε Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο να εξασφαλίσουμε ότι στα κράτη-μέλη και σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης θα υπάρχει μια διατύπωση η οποία δεν θα είναι τεχνική, δεν θα είναι ιδιαίτερα επιστημονική, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Φτάνει. Ε, Ευχαριστώ. Γιωχάνες. Έχουμε κάποια λεπτά για τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Μάρκους Πίπερ. Α, προηγουμένως, ο κύριος Μικολάσετς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας. Και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Ρόσπαχερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας διαβεβαίωσω ως προς το... Πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση και όπως δήλωσα στην αρχή, είμαι ανοιχτός. Θα δεχτώ τα σχόλια και τις υποδείξεις σας. Αλλά το χρονοδιάγραμμα για το έργο που έχουμε μπροστά μα δεν το είδα. Απλώ να σα πω ότι η προθεσμία για την υποβολή και την κατάθεση τροπολογιών είναι η Τετάρτη Φεβρουαρίου. 4 Φεβρουαρίου πιο συγκεκριμένα. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν τροπολογιε Προσωπικώ θα καταθέσω και εγώ τι δικε μου τροπολογιε γιατί οπω θα ακούσατε η έκθεση αυτή είναι σχετικώ περιορισμένη τον αριθμό των λέξεων 3.500 λέξεις έπρεπε να έχει. Προσωπικώς λοιπόν θα καταθέσω και εγώ κάποιες τροπολογίες γιατί νομίζω ότι θα βελτιώσει αυτό το κείμενο. Σας καλώ όμως αγαπητοί συνάδελφοι να καταθέσετε τις δικές σας τροπολογίες και είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε συνεννόηση, σημεία συνεννόηση, παιδεία συνεννόησης και συμβιβασμού. Και είμαι διατεθειμένος να λάβω υπόψη μου όλες τις ποιοτικέ τροπολογίες που θα καταθέσετε και θα υποβάλλετε. Οι τροπολογίες αυτές θα μεταφραστούν στις 21 Φεβρουαρίου. Η υιοθέτηση στην Επιτροπή Ρέτζη έχει προγραμματιστεί για την 21η-22η μαρτιου Και μιας και, επειδή μάλλον έχουμε πολλά νομοθετικά κείμενα προς υιοθέτηση στην Ολομέλεια του Απριλίου, το κείμενο αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει στην Ολομέλεια του μηνός Μαΐου στο Στρασβούργο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ Μυρόσλαβ. Έκανε το έργο μου. Δεν χρειάζεται να παραλάβω όλα αυτά τα πράγματα. Πράγματα τα οποία πρέπει να τα πει η Προεδρία. Αλλά να σε διορθώσω, διότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 3 Φεβρουαρίου, 6 το απόγευμα. Τώρα, Έχουμε δύο λεπτά ανά ομιλητή, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε το σκιώδη εισηγητή, από θα ήθελα να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από του σκιώδη εισηγητέ και κατόπιν ο κ. Μάρκο Πίπερ. Η Ουλρίκα Μάνερ είναι η πρώτη που θα λάβει το λόγο. Εκτό αν δεν θέλει να λάβει το λόγο. Πείτε, πε το μου, αν δεν θέλει να λάβει το λόγο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική πραγματικά δουλειά του. Και έχω βεβαίω κάποια πολύ σύντομα σχόλια τα οποία θα ήθελα να διατυπώσω. Διότι μου φαίνεται ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντε ελήφθησαν υπόψη σε αυτό το σχέδιο γνώμη. Και ευχαριστώ τον κύριο Ροσμπάχερ για την παρουσίασή του, την οποία βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Εδώ, όταν γίνεται λόγο και όπου γίνεται λόγο για την πολιτική συνοχή, και τα ταμεία για την περιφερειακή πολιτική και όλα αυτά, εκθέσεις του είδους αυτού είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και βλέπω εδώ ότι ελήφθησαν δεόντως υπόψη, νομίζω, τα βασικά και τα βασικότερα στοιχεία, τα οποία μας επιτρέπουν να σπρώξουμε τα πράγματα, να ενισχύσουμε δηλαδή την πολιτική μας, να σπρώξουμε τα πράγματα δηλαδή προς την κατεύθυνση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία του είδους αυτού, όταν έχουμε συζητήσεις πάνω στα θέματα αυτά. Πρώτα απ' όλα, Μια ερώτηση θα ήθελα να υποβάλω όσον αφορά τις εθνικές εκθέσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι εκθέσεις και να υποβληθούν αυτές οι εκθέσεις, αλλά οι εκθέσεις αυτές πρέπει κατά τη γνώμη μου να παρουσιάζουν και τις περισσότερες ομοιότητες για να μπορούν να θέλετε να συγκριθούν η μία με την άλλη. Να υπάρχει δυνατότητα σύγκριση δηλαδή μεταξύ αυτών. Και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε και σαφέστερα αποτελέσματα ως προς την ερμηνεία τους. Διότι όπω πολύ σωστά είπε ο κύριο Σίγητης, δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα πάντα. Πρέπει να, αυτό να το λάβουμε υπόψη στις εθνικέ εκθέσει και να λαμβάνεται υπόψη. Επίση, το ζήτημα της ενίσχυσης τη περιφερειακή πολιτική. Ο Συγητή αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και βεβαίω αυτό σχετίζεται και με άλλε πολιτικέ. Πρέπει και χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη συνεργασία με άλλου τομείς πολιτική, την έρευνα και την ανάπτυξη Φερρυπίν διότι νομίζω ότι στην περιφερειακή πολιτική θα μπορούσαμε και μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλους τομείς όπως αυτόν που ανέφερα προηγουμένως. Χρειάζεται συνεπώς συνεργασία διατομεακή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να πούμε να άρουμε και να καταστρέψουμε αν θέλετε τους φραγμούς που υπάρχουν μεταξύ αυτών των τομέων τη σήμερα ημέρα. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων αν θέλετε ποικίλει Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία είναι πιο αποτελεσματικά και άλλα λιγότερο. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να διδαχθούμε από τις διαδικασίες αυτές και να πάρουμε δηλαδή και να αφομοιώσουμε και να απορροφήσουμε θέλετε, τα απαραίτητα θέλετε, διδάγματα. Τώρα και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφή αποτελέσματα. Σε όλα τα έργα δηλαδή τα οποία υλοποιούνται διότι τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν είναι και τόσο σαφή. Αν είχαμε καλύτερα αποτελέσματα θα μπορούσαμε να δούμε καλύτερα πού σημειώθηκε η επιτυχία και να ενισχύσουμε βεβαίω τη σχετική πολιτική. Η επιλογή των έργων επίσης. Αυτό επισημαίνεται στην έκθεση. Αν δεν υπάρχει σαφής προτεραιότητα, τότε τα προγράμματα δεν εξυπηρετούν κανένα με κανένα σκοπό. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που θα ήθελα να διατυπώσω. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι πραγματικά μια έκθεση ποιότητος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάτεμπερκ, εν συνεχεία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ακόμα και αν δεν έχουμε πολύ χρόνο για να λάβουμε το λόγο, θέλω να ευχαριστήσω τον Αυστριακό συναδελφό μου για την έκθεση την οποία παρουσίασε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγήτη. Και επίσης ήταν πάρα πολύ επακριβής και ενδιαφέρουσα η έκθεση και ακόμα και αν έρθουν τροπολογίες από τη δική μας ε, παράταξη, εγώ θέλω να τονίσω ότι κατά την άποψή μου είναι μια πολύ καλή έκθεση η οποία ε, εστιάζει στα ουσιώδη στοιχεία και γι' αυτό εγώ χαίρομαι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν ασχολείται με λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να είναι και άχρηστες αλλά εστιάζει πάρα πολύ στο, στα βασικά θέματα. Από την οπτική γωνία και πάλι της Αυστρίας νομίζω ότι είναι πολύ καλά αυτά τα οποία αναφέρονται και προφανώς αυτά που είπατε θα χρειαζόταν ίσως περισσότερο χρόνο για συζήτηση αλλά με ενδιέφερε πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία για να θεσπίσει κατευθύνσεις και ότι δεν πρόκειται μονάχα για την ε, χρήση εργαλείων τα οποία δεν ε, βοηθούν να προχωρήσουμε. πολλέ φορέ. υπάρχουν βέβαια διαδικασίε, οι οποίε είναι χρονοβόρες, όπω παραδείγματο χάρη η συλλογή των πληροφοριών που είναι απαραίτητε και είναι απαραίτητε και οι πολιτικέ συζητήσει, οι οποίε θα καταλήξουν σε μια πιο ενδελεχή μορφή σχεδίαση, Αλλά παράλληλα πρέπει να υπάρχουν και εργαλεία τα οποία θα μα βοηθήσουν να κάνουμε γρήγορε αλλαγέ κατευθύνσεων, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Συνάδελφοι, παρακαλώ να είστε όσο πιο σύντομοι γίνεται γιατί θα πρέπει να ακούσουμε και την Ουγγρική Προεδρία. Οι επόμενοι ομιλητέ. Τα δύο λεπτά που έχετε στη διάθεση μπορείτε να τα μοιράσετε, παρακαλώ. Πάρα πολύ γρήγορα. Δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Είναι σαφές ότι εδώ μιλάμε για εθνικά προγράμματα πλαισίου. Εδώ το πρόβλημα είναι πώς κρίνω αν ένα πρόγραμμα είναι επιτυχές άμα δεν γνωρίζω το γενικό στρατηγικό πλαίσιο και εξάλλου θα πρέπει να έχουμε και κάποια συζήτηση για το outcome, για την τελική απόλυξη ενός προγράμματος και όχι μονάχα για το γενικό πλαίσιο. Επίσης, θα έπρεπε να υπάρξει και μείωση της γραφειοκρατίας, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Και ήθελα να πω Μίκαελ ότι μία ε, προσπάθεια η οποία έχει σαν στόχο το αποτέλεσμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχουν οι σωστές δομές επιτοπίως. Αυτό λοιπόν πρέπει ήδη σε επίπεδο προγράμματος να γίνεται και να συνδέεται με τις εθνικές ε, συνθήκες και τα εθνικά προγράμματα. Το δεύτερο που φάνηκε από την έκθεση αυτή επίσης είναι ότι όπως είπατε η εταιρική σχέση και η συνεργασία μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο, ιδίως όταν πρόκειται για καινοτόμε ενέργειες. Ένα, αυτό ίσως δεν αντανακλάται αρκετά στην έκθεση του κυρίου Μικολάσιτς. Ένα τρίτο σημείο ε, ήταν ότι ήταν ενδιαφέρον να μπορέσουμε να εξετάσουμε και την ε, σωστή χρήση των εργαλείων αυτών μέσα στο πλαίσιό τους. Αυτό είναι κάτι που το υποστήριξαν τα περισσότερα κατημέλη και οι περισσότεροι βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε όμως ότι το κάθε ταμείο πολλές φορές έχει τους δικούς τους κανόνες και επομένως αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε επικαλύψεις. Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε. Μήπως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε περισσότερο στα ζητήματα αυτά τα οποία είναι ολοκληρωμένου χαρακτήρα να εστιάζει το Ταμείο Συνοχή στην προσπάθειά του, ενώ υπάρχει η τάση να κόβεται σε φέτε και να εξυπηρετεί διάφορου τομεί. Πιστεύω ότι αυτοί οι στόχοι οι οποίοι τίθενται ανατομέα δεν θα πρέπει να διαταράσουν τη γενικότερη στόχευση η οποία γίνεται σε ολοκληρωμένο επίπεδο. Αυτά και ο Μιχαήλ θα συνεχίσει. Thank you. you have to... Κύριε να είστε σύντομος παρακαλώ. Υπάρχουν, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποια σημεία στο σχέδιο ε, έκθεσης του κύριου Μικολάση. Ε, γενικά είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Τα δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω πολύ σύντομα στο εισαγωγικό κεφάλαιο, στην παράγραφο 3 που γίνεται αναφορά για την ε, διαφάνεια, στην ανάθεση των κονδυλίων ως βασική προϋπόθεση στην επίτευξη των συνολικών στόχων της πολιτικής συνοχής και ως ε, τέτοια πρέπει να ενισχυθεί. Προφανώς συμφωνούμε, όμως ε, ήδη παρακάτω στην παράγραφο 17 αναφέρεται πως είναι αδύνατο να έχουμε μια συνολική εικόνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς μόλις 19 χώρες έχουν δώσει τους βασικούς δείκτες που απαιτούνται για να γίνει η σύγκριση. Ενώ και στην παράγραφο 18 ζητάμε από την Κομισιόν να ενισχύσει τη συνεκτικότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνει. Διαπιστώνουμε λοιπόν ένα κενό διαφάνειας, ένα έλλειμμα δεδομένων που σωστά εντοπίζεται. Πρέπει όμως να είμαστε ξεκάθαροι ε, και ενωμένες στην ανάγκη για διάχυση και αξιοποίηση των απαραίτητων αυτών στοιχείων. Στην έκθεση, στο κεφάλαιο της εφαρμογής, στην παράγραφο 6 γίνεται λόγος για ελλειπείς δείκτες αποτελεσμάτων και δεδομένων για όλα τα κράτη μαζί. Ε, θα πρότεινα λοιπόν να υπάρχουν μια σειρά από για τις χώρες που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, για παράδειγμα θετική δημοσιότητα και προβολή. Για τις χώρες όμως που υστερούν θα πρέπει να σκύψουμε με προσοχή και αφενός να βοηθήσουμε, αφετέρου να στυλιτεύσουμε τα όποια φαινόμενα αδιαφάνειας και αδράνειας, να είμαστε αυστηροί εκεί που χρειάζεται. Το άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ είναι στην παράγραφο 7, όπου γίνεται λόγος για καθυστερήσεις στην επιλογή έργων στρατηγικής σημασίας, όπως είναι διάφορα ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα, τα έργα ψηφιακής οικονομίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, ο σιδηρόδρομος και άλλα. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να αναλάβουν δράση και να προχωρήσουν με γρογούς ρυθμούς στις αναγκαίες εκείνες δράσεις που θα φέρουν υψηλότερη απορρόφηση. Θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Επιτροπή. Δεν μπορεί οι συνολικές πιστώσει των επιλεγέντων έργων να έχουν μέσο όρο 27,1% εννιά χώρες να εμφανίζουν πρόοδο με ποστά επιλογής άνω του 40% ενώ τέσσερα κράτη-μέλη να είναι κάτω του 20%. Για ποια συνοχή, πολιτική συνοχής μιλάμε λοιπόν, δύο και τριών ταχυτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ο κύριος Paní dámy Κυρίε και κύριοι, και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για αυτή την έκθεση. Είναι η πρώτη τέτοια ανάλυση των ε, εφαρμογών προγραμμάτων αυτού του είδους σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Είναι κρίμα που δεν έχουμε όλους τους δείκτες και όλα τα αποτελέσματα, τα outcomes από όλα τα κράτη-μέλη. Επομένως αυτό κάπως μειώνει την αξία της, της ανάλυσης αυτής. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν διορθώσει γιατί αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δώσει ακόμα τα στοιχεία θα πρέπει να κολλαστούν και θα πρέπει να τους πούμε με τρόπο αυστηρό ότι πρέπει να μας δώσουν αυτά τα στοιχεία. Πολλές φορές έχουν καθυστερήσει αυτά τα προγράμματα λόγω της ε, βραδίας εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Πολλές φορές δεν υπήρχε το απαραίτητο έμψυχο υλικό. Και θέλω εδώ να αναφέρω ένα ιδιαίτερο τομέα, στον οποίο έχω ενδιαφέρον, πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τον κατακυρματισμό των προσπαθειών σε διάφορες περιοχές πολιτικής. Δεν αφορά αυτό μόνο το Περιφερειακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια σύνδεση προς το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης επίσης. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν μιλάμε για την Ήπεθρο. και το αγροτικό χώρο. Όλα αυτά λοιπόν, όλοι οι κανόνες θα πρέπει να απλοποιηθούν αν θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτόν τον τομέα, γιατί πολλές φορές υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις οι οποίες επισυμβαίνουν λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας. Ευχαριστώ και πάλι τον συγητή και θα κατεθέσω κάποιες τροπολογίες. Ο Μάρκους. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πάρα πολύ. Σύντομα και εγώ θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι και οι δύο παρουσιάσεις του εισηγητή και του κυρίου Ροσπέργκερ ήταν ιδιαίτερα θετικές και πιστικές. Τι έχουμε μάθει από όλα αυτά. Ότι ο προσδιορισμός της ε, ε, Λισαβόνα, 63 δισεκατομμύρια, λειτουργήσε πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι η διαρθρωτική μα πολιτική έχει λειτουργήσει πολύ καλά και έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει και τα συγκυριακά προγράμματα, δηλαδή μα δίνει ένα αρκετά ευέλικτο πλαίσιο. Μάθαμε ότι υπήρξε μια σχετικά υψηλή απορρόφηση σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ω εκ τούτου μπορώ να εκφράσω την άποψη ότι το σύστημά μα και η στοχοθεσία και η δομή του προϋπολογισμού έχουν αποδείξει την αξία του και δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την στρατηγική Ευρώπη 2020 με τελείω νέε δομέ. Αυτό είναι ένα δίδαγμα το οποίο έχουμε αποκομίσει. Εγώ λυπάμαι βέβαια για τι καθυστερήσει οι οποίες συνέβησαν. αλλά το θέμα είναι πώ μπορούμε να τι απο... αποτρέψουμε τι καθυστερήσει στο μέλλον με μια απλοποίηση των κανόνων του Περιφερειακού Ταμείου, ώστε να μην είναι τόσο δύσκολη η εφαρμογή του στην πράξη. Και επίσης γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε κάποιους κεντρικούς δείκτες οι οποίες μπορούν να καταδείξουν με καλύτερο τρόπο την ε, πρόοδο και όταν βρισκόμαστε σε, στη σύγχρονη εποχή με τον ψηφιακό ε, χρόνο μπορούμε να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες χρησιμοποιώντας μοντέρνες μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και στον κύριο Ροσμπέργκερ, νομίζω ότι, Ροσμπάχερ, νομίζω ότι δείξατε ότι μπορείτε να προσαρμοστείτε σε αυτό το χρονικό ε, πλαίσιο με τις προσπάθειες που καταβάλλετε. Φανίστε, Ρόι. Μια ερώτηση. Βάση και δυνάμει αυτής της τόσο καλής εκθέσεως. Αν δείτε το ερώτημα που έθεσε ο Μάρκος, κατά την εξή έννοια, ότι έχουμε τα διάφορα ταμεία. Έχουμε το Περιφερειακό Ταμείο, το Αναπτυξιακό Ταμείο Ανάπτυξη, το Ταμείο Συνοχή, το Κοινωνικό Ταμείο και πάει λέγοντα. Και αν, εάν λέω, αυτή τη στιγμή τη μετάβαση, τη μεταβατική περίοδο δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτά θα πρέπει να τα συνενώσουμε, τα ταμεία δηλαδή, ή πιστεύετε είναι η γνώμη σας για να θέλετε τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα. Διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά καλύτερο συντονισμό σε αυτόν. Και η διαφοροποίηση των στόχων που υπάρχει πριν στην περιφερειακή πολιτική, στο Ταμείο Συνοχής και η σχέση, αν θέλετε, με άλλα εργαλεία. Θα ήθελα, αν θέλετε, αυτά τα πράγματα να ληφθούν υπόψη να θέλετε στην ε, συζήτηση. Ο κύριος Μάγερ, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ροσμπάχερ. Τρία θέματα θέλω να θέσω, τα οποία έχουν πρακτικό χαρακτήρα. Έχουμε συμφωνία για την ε, σημασία αυτής της στρατηγικής και αυτό είναι κάτι το θα είναι σημαντικό και σε μελλοντικέ συζητήσεις, να δούμε πώς θα υπάρχει δεσμευτικότητα για την ε, παροχή αυτής της ε, Εκθέσεω, γιατί μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε μεταγενέστερες συζητήσει. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση της ε, Αυστρίας. Στην περίπτωση της Αυστρίας υπήρχαν και επικρίσεις από το ελεκτικό συνέδριο για τη χρήση των πόρων. Αυτό είναι θέμα το οποίο και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα των πόρων οι οποίοι δεν έχουν απορροφηθεί και οι οποίοι συσσωρεύονται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή θα πρέπει να χαθούν. Και η τρίτη πλευρά, κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι το γεγονός 25% της εκτέλεσης έγινε στην περιοχή της ε, πρωτεύουσας μονάχα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά είναι συνολικά πόσα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική εφαρμογή στο μέλλον, ώστε να υπάρχει και περισσότερη υποστήριξη στι περιφερειακέ πρωτεύουσε και στον χώρο τη υπαίθρου. Μήπω χρειάζεται να υπάρξει διαφορα... διαφορετική αντιμετώπιση στο σχεδιασμό μα. Ευχαριστώ, ο κ. Σκέλη. Θα είμαι και εγώ σύντομο, σα το υπόσχομαι, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον φίλο και συνάδελφο, τον κύριο Μιλάσεκ, για το... την πολύ καλή δουλειά του. Κάτι το οποίο ανέφερε και το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να επισημάνουμε αυτή την πρακτική. Και λέγοντα αυτά, αρκετά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό ή να δώσουμε απλά παραδείγματα. Και ο κύριο Ροσμπάκερ ε, ήρθε παρουσιάζοντα το αυστριακό παράδειγμα, το οποίο μα ενέπνευσε πολύ και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά που είπε. Να επισημάνω ένα μόνο εξ αυτών. Είπε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο όλοι πλέον γνωρίζουμε χρησιμοποίησε την εξή φράση. Over academic στο report, δηλαδή πολλές φορές χρειάζεται έξι μήνες για να ετοιμαστεί αυτή η έκθεση. Μεταξύ δηλαδή της υποβολής των εκθέσεων και των αιτήσεων περνάει πολλής χρόνος. Πολλές δαπάνες, διοικητικές δαπάνες, τα οποία αν θέλετε σε τελική ανάλυση δεν προσφέρουν και κανένα όφελος αν θέλετε και δεν δημιουργούν πλέον εκτίματα δηλαδή για το χρηματοδοτούμενο αυτό έργο. Αν όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε ένα μήνα, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι δεν πάει καλά. Και πρέπει οπωσδήποτε και σύμφωνα με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Τόσο σε αφορά τι αιτήσει, να αφορά επίση και την υποβολή των εκθέσεων. Και να θέσουμε, αν θέλετε, στόχου χρηματοδότηση στα έργα αυτά που δημιουργούν, αν θέλετε, αυτά τα οικονομικά ωφέλη και πλεονεκτήματα. Ευχαριστώ και πάλι, πάντω. Ευχαριστώ πολύ, Σον. Επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να Λαμβάνω το λόγο προκειμένου να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Μύροσλαβ και να πω ότι το έγγραφο είναι ιδιαίτερα θετικό και περιέχει συμπεράσματα τα οποία καταλήξει η ίδια η Επιτροπή όταν ε, συνόψισε τις ε, εθνικές ε, εκθέσεις συνοχής για μια ολοκληρωμένη πολιτική συνοχής και να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό και να υπάρξει μια εναρμονισμένη ανάπτυξη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, οι οποίες θέλουν να τονίσουν τις ε, θετική, σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτική συνοχή, στην ε, πολιτική έρευνας, παιδείας, υγείας και επιχειρήσεων. Χρειάζεται λοιπόν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά τα ζητήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις ε, καθαρές ε, συγκοινωνίες, καθαρά μέσα μεταφοράς κλπ. Επίσης να πω κάτι για τις ε, περιοχές που βρίσκονται σε δύσκολη, σε θέση όπως οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές και στην περίπτωση της Ισπανίας, στην Θέουτα και της Μελίδια, που είναι παραμεθόρες περιοχές διαφορετικές από ό,τι στην, ε, έχουμε συστήσει στην Ευρώπη που αποτελούν τα σύνορα με την ε, Αφρικανική Ήπειρο κάτω από συγκεκριμένε και ιδιαίτερε προϋποθέσεις. Χρειάζεται λοιπόν να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα αυτή. Είμαι μέλος της Επιτροπής ε, ε, ε, ε Περιφερειακής Επιτροπή και τη Επιτροπής Γυναικών και φαίνεται η Επιτροπή Γυναικών θα υιοθετήσει κάποιε τροπολογίες προκειμένου να προωθήσει το ζήτημα του φύλου αναφορικά με τι πολιτικέ ε, κατάρτιση και για να προωθήσει μέσω αυτής την πολιτική ισότητα των φύλων. Να ξέρετε ότι θέλαμε να τις υποστηρίξετε και εσείς προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας στην Επιτροπή Γυναικών. Τελειώσατε τα σχόλια συνάδελφοι. Τότε θα μπορούσα να είμαι ιδιαίτερα γενναιόδορη και να δώσω ένα λεπτό επιπλέον στον Ιωάννης και στον ε, Νίκολας. Ποιος επιθυμεί... Κύριε Αγκουράκη, δεν είχαμε σημειώσει ότι επιθυμούσε να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Είτε για τη δυνατότητα να σε ευχηθώ καλή χρονιά, Πρόεδρε. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, η έκθεση, η έκθεση ε, η έκθεση αναφέρεται όντως στα προγράμματα και στον τρόπο υλοποίησής τους. Η απορία που έχω εγώ είναι η εξής. Επειδή κάνει μια ε, αναφορά και ο εισηγητής, ε, αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι το σημείο 10 που εκφράζει τη λύπη του για το ότι δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά την κατάσταση των ανισοτήτων το 2009. Δεύτερο εισηγητής, θα είναι σοβαρό πρόβλημα. Αυτό σε συνδυασμό με το σημείο 17, πολύ σωστά η έκφραση εκφράζει τη λύπη του για το ότι υπάρχουν στοιχεία μόνον από 19 κράτη-μέλη. Ε, το θέμα που θέτω εγώ στον εισηγητή είναι το εξή, χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία της έκθεσης κτλ. Από τα στοιχεία που είχε εκείνο υπόψη του, δεν θα μπορούσε να μας δώσει μια εικόνα εάν έχουμε σύγκληση ή απόκληση. Και το ίδιο ερώτημα θα ήθελα να θέσω στον κύριο Ροσμπάχερ όσον αφορά τις αυστριακές περιοχές. Μας είπε ότι κάποιες είναι στο στόχο της σύγκλησης και κάποιες είναι στο, στόχο, στο στόχο της ανταγωνιστικότητας. Το ερώτημα που έχω εγώ είναι στην Αυστρία, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αυστρία οι περιοχές της σύγκλησης συγκλίνανε με αυτές της ανταγωνιστικότητας. Με ποιον συγκλίνανε και σε τι βαθμό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μύροσλαφ, σε παρακαλώ να είσαι όσο πιο σύντομο γίνεται. Ο Μύροσλαφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα περιοριστώ στι ευχαριστίε μου προ του συναδέλφου, όλου του συναδέλφου που τοποθετήθηκαν για τα σχόλια, για την εκτίμηση που εξέφρασαν και τις ε, ιδέες τους που ήταν εμπνευστικέ, όπως θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω. Απλώς και για να μην απαντήσω σε όλους σας, σημείωσα, κατέγραψα ότι ορισμένα κράτη-μέλη που έπρεπε να αναφέρω ότι υπολείπονται εναντί των ε, υπολείπων δηλαδή, εντωμεταξύ βελτίωσαν τη θέση του. Η χώρα μου, Σλοβακία Φερρυπίν, άλλαξε κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση τώρα πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι προηγούμενη σε όλα τα θέματα δηλαδή που άπτονται αν θέλετε της περιφερειακής πολιτικής και της απορρόφησης πόρων και κονδυλίων. Βεβαίω έγινε ζήτημα συγκρίσιμων δεδομένων. Είναι ζήτημα μεθοδολογικό αυτό και έπρεπε να κάνω την διαπίστωση στην εξή. Ορισμένα κράτη-μέλη απήντησαν σε ερωτήσει ρωματολογίου διαφορετική χρονική στιγμή από ό,τι τα υπόλοιπα. Επομένω η σύγκριση ήταν κάπω δυσχερέστερη, πιο δύσκολη αλλά νομίζω ότι θα μπορούσα να πω ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ως προς το μέλλον. Γιατί οι συνάδελφοι θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν τα διάφορα αυτά κονδύλια μέχρι το 2015. Διότι δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση, αν θέλετε, της περίοδου αυτής, το 2014 δηλαδή, μένουν άλλα δύο χρόνια. Μένουν άλλα δύο χρόνια. Άρα, μέχρι το 2015, πολλά κράτη-μέλη, πιστεύω, και αυτό αναφέρεται στην έκθεση, θα έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι τώρα. Και καλό όλους σας και πάλι να συζητήσετε μαζί μου ή να καταθέσετε τις τροπολογίες σας γιατί νομίζω ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε τελικά να φτιάξουμε αν θέλετε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Γιωχάννη. Μπορείς να θέλετε να σχολιάσει και εσύ συντομία, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσετε να λάβω το λόγο εδώ και ίσως ένα-δυο σημεία μονάχα. Το θέμα της χρόνισης των εκθέσεων είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί διαμακρών. Είμαι στη διάθεσή σας στο διάδρομο ή σε κάποια άλλη χρονική στιγμή, γιατί φοβάμαι ότι αυτό το θέμα θα καταδαπανούσε πάρα πολύ χρόνο. Δεν θέλω να καθυστερήσω τη μέση διαταξή σας. Είμαι βεβαία ότι ο κύριος Ροσμπάχερ είναι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση και μάλιστα και από τη Βιέννη. Αν θέλετε να δείτε, να μελετήσετε τις βέλτιστες πρακτικές που αξιοποίησε και χρησιμοποίησε η Αυστρία. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλους και η, όπως σας είπα 6 δολαρίου σε 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών σας, υποβολή των τροπολογιών σας. Γι' αυτό λοιπόν ας είσαστε, παρακαλώ να είστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Ο Όλτεχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για αυτά που έκανε η κυρία Σμιθ στην ε, Επιτροπή Πολιτισμού που ήταν αρμόδια για αυτή την έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω επίσης και την συνάδελφό μας την κυρία Σμόλκοβα για τη συνεργασία της. Ήμουνα σε επαφή μαζί της και με άλλους που ασχολήθηκαν με αυτή την έκθεση. Η γνωμοδότησή μας βασίζεται στην ε, Διαβούλευση με συναδέλφους από τοπικές και περιφερειακές αρχές. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η έκθεση της Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συζήτησε την έκθεση αυτή το φθινόπωρο. Ήταν η κυρία Σικοβάτσικα από τη Νότια Μοραβία που, που αντιμετώπισε αυτό το θέμα. Και είναι πολλά τα στοιχεία που μπορέσαμε να βγάλουμε από τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν της ε, Πράσινης Βίβλου. Ελπίζω ότι έχετε την ε, γνωμοδότηση αυτή ενώπιόν σας. Ένα-δύο πράγματα μόνο θέλω να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, εμείς θα πρέπει να αναλύσουμε και τα αποτελέσματα της κατανομής των, ε, από την πλευρά της Κομισιόν στις, στους διάφορους οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τα αποτελέσματα αυτής της κατανομής ώστε να έχουμε δυνατότητες να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη. Θα πρέπει να εμπλέξουμε περισσότερο ιδιωτικό κεφάλαιο, να έχουμε περισσότερες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα αυτό, ώστε να προσελκύσουμε και περισσότερες βιώσιμες επενδύσεις. Και να μην είναι απλώς όλα αυτά τα θέματα ένα ζήτημα απορρόφησης κονδυλίων Πιστεύω ότι θα υποστηρίξετε και εσείς αυτή την αντιμετώπιση, γιατί η Πράσινη Βίβλος είναι απλώς η απαρχή μιας διαδικασίας διαβουλεύσεων και χάραξης πολιτικής. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε άκαμπτους κανονισμούς και κανόνες. Αντίθετα, <clears throat> θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Και εν κατακλείδη, <clears throat> θα υποβάλω και ο ίδιος κάποιες τροπολογίες για το κείμενο το οποίο έχετε ενώπιόν σα και ο κύριος Μικολάσικα έκανε το ίδιο και έχουμε φυσικά προβλήματα με το μήκος της γνωμοδότησης που είναι περιορισμένη και ίσως με τροπολογίες και αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε μερικά ακόμα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Εμάς μας ενδιαφέρει η πρωτοβουλία για την, της, για την Ευρώπη της καινοτομίας και την ψηφιακή ατζέντα πρέπει να, να υπογραμμίσουμε τη σημασία των τελεχνολογιών ε, επικοινωνιών και πληροφορικής για την υποστήριξη της βιομηχανίας καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως η συλλογή και η ψηφιοποίηση στοιχείων που μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες ως ε, εξέχοντα παραδείγματα ευρωπαϊκής συνεργασίας που με την υποστήριξη του πολιτισμού επιτρέπουν την αναζωογόνηση των πολλών πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούν και βέλτιστες πρακτικές οι οποίες μπορούν να μεταλαμπαδευτούν μεταξύ κρατών μελών. Τέλος, θέλω να τονίσω την ε, σημασία της λεγόμενης αδελφοποίησης πόλεων και δήμων. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πάντα στον τομέα αυτό και θέλω να κάνω μια έκκληση στην Κομισιόν μαζί με τις ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών να συνενώσουν τις προσπάθειές τους και να βρουν καλύτερο τρόπο να αναπτυχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Έχω σταθεί και εγώ δημοτικός άρχον και γνωρίζω πόσο μεγάλη είναι η σημασία των αδελφοποίησεων για την πολιτιστική συνεργασία. Αυτά λοιπόν και περιμένω και τα δικά σας σχόλια, αγαπητοί συνάδελφοι και τις ιδέες για τροπολογίες. Ο κύριος Κέλλη. Δύο λεπτά παρακαλώ. Δείξτε μας ότι μπορείτε κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό και καλό κάνουμε που δίνουμε προσοχή στην πολιτιστική, αν θέλετε, και δημιουργικές βιομηχανίες γιατί παρουσιάζουν πολύ δυναμικό στην Ευρώπη και πολλοί δεν το αναγνωρίζουν αυτό. Δεν αναγνωρίζουν δηλαδή, τη συσφορά και τη συνδρομή του. Το 2,6% δηλαδή του ΑΕΠ. Και ευθύνουν δηλαδή για 5 εκατομμύρια θέσει εργασία. Αλλά δεν βρίσκονται, αν θέλετε, στον κορμό, τη βασική οικονομική δραστηριότητα. Και νομίζω ότι αυτή η γνωμοδότηση θα βοηθήσει να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Επίση υπάρχουν και κάποιε επιπτώσει στον τουρισμό. Και αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στην πράσινη βίβλο. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί. Τώρα βεβαίως κάποια από τα διορθωτικά ταμεία χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αναπτυχθούν κάποιες από τις υποδομές. Υποδομές που απαιτούν αυτή η κλάδη. Δηλαδή τέτοιου γκαλερί, έργων τέχνης κτλ. Δημόσιες αν θέλετε πινακοθήκες κτλ. Πρέπει όλα αυτά να τα ξαναδούμε και ως κομμάτι αν θέλετε στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 είναι να φτιάξουμε, θέλετε, τις ευρυζωνικές ε, υψηλής ταχύτητος σε όλη την Ευρώπη, τις διασυνδέσεις αυτές. Διότι η πολιτική βιομηχανία, αν δεν έχει, αν θέλετε, το κόλλημα, αν θέλετε, της θέσεως, αν θέλετε, και του τόπου. Γιατί μόλις υπάρχει η τεχνολογία, η μουσική, οι ταινίε του κινηματογράφου δηλαδή, μπορούν να προβληθούν παντού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να τονίσουμε και να επισημάνουμε και να αναπτύξουμε όχι μόνο όσον αφορά θέλετε τις κοινωνικές του επιπτώσεις, αλλά και τα οικονομικά ωφέλη που μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη των βιομηχανιών αυτών και των κλάδων αυτών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και που θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Κάτι άλλο τώρα θα πρέπει να δώσουμε, αν θέλετε, και να βρούμε, αν θέλετε, και να διαθέσουμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Γιατί πολύ συχνά οι κλάδοι αυτοί έχουν, αν θέλετε, κάποια υγιή επιχειρηματικά σχέδια Όπω θεωρούνται δηλαδή από τις τράπεζες και τους άλλους πιστοτικού φορείς. Και αν μπορούν να αντλήσουν κάποια χρήματα, αυτό θα τους βοηθήσει να βρουν, αν θέλετε, και να φέρουν με το μέρο του, αν θέλετε, και άλλους εταίρου, συνεταίρου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτό και στην πρόσφατη απόφαση που ελήφθη για να διατεθούν, αν θέλετε, αυτά τα εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη μορφή δανείων και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε, διότι ο αντίκτυπο θα είναι τεράστιο και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκλειδώσουμε, αν θέλετε, το δυναμικό, αν θέλετε, τη δημιουργική βιομηχανία και να αυξηθεί ο αριθμό των απασχολουμένων στου κλάδου αυτού. Πολύ περισσότερο μελλοντικά. Και να εγγυηθούμε βεβαίω και την πολιτιστική ποικιλομορφία τη Ευρώπη και τη διατήρηση πολλών πολιτικών στοιχείων σε πολλά σημεία τη Ευρώπη. Είτε είναι μεμονωμένε και απομονωμένε περιοχέ, ή αν θέλετε οι μεγάλε πόλει, αν θέλετε και αστικά κέντρα. Αυτά είχα να πω και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι σκιώδει συγητές που θέλουν να λάβουν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγα λόγια να πω. Η ομάδα μας ε, είναι υπέρ αυτή τη ε, συμπερίληψη ε, του κλάδου ε, πολιτισμού και της δημιουργικότητας για την περιφερειακή ανάπτυξη και για μα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον που το ζήτημα αυτό έρχεται ενώπιον του Κοινοβουλίου. Να πω επίσης προς τον εισηγητή ότι το σύνολο των σημείων που φύγει είναι σημεία τα οποία μπορούμε να στηρίξουμε, δεν έχουμε καμία ένσταση να κάνουμε, αλλά μία προσθήκη η πρώτη ύλη αυτή τη ανάπτυξη είναι η πολιτισμική διαφορά και επικοινωνία της Ευρώπης. Υπάρχουν ε, σήμερα κάποιε ε, πολιτισμοί που απειλούνται με εξαφάνιση, κινδυνεύουν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η προβληματική χρειάζεται να τονιστεί περαιτέρω στο κείμενο. Πρέπει να θυγεί διότι ε, αν χάσουμε ένα τμήμα του της Ευρώπης σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και μία, ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η μεγάλη ποικιλομορφία ακριβώ των πολιτιστικών στοιχείων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και μας διαφοροποιεί από τους άλλους και δεν μπορούμε να λέμε ότι αφενός θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις ε, αυτούς τους κλάδους ε, πολιτισμού και δημιουργικότητας, αλλά παράλληλα να μην κάνουμε τίποτα για να τους βοηθήσουμε θα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαι βέβαια η κυρία Σμόλκοβα, αλλά η κυρία Σμόλκοβα μου ζήτησε να ε, μεταφέρω τις ε, απόψεις της, γιατί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να έρθει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδίτησής του. Βλέπουμε ότι μέσω της πράσινης βίβλου ζητείται να παίξει ένα ρόλο η κουλτούρα και να αναγνωριστεί ως εργαλείο για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι οι δυνατότητες απασχόλησης οι οποίες παρέχονται από την κουλτούρα, αλλά συγχρόνως και το θέμα της ανταγωνιστικότητας που μπορεί να βελτιωθεί μέσω του τομέα του πολιτισμού. Τονίσατε ότι πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο ακριβώς πώς μπορεί να υπάρχει καλύτερη κατανομή των χρηματοδοτήσεων. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στους ε, φορείς τους πολιτιστικούς επιχειρήσεις στον τομέα αυτό να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση αυτή και πέραν των επιδοτήσεων, πέραν των δημοσίων κονδυλίων, να υπάρχει δυνατότητα να προσελκύσουν και ιδιωτικούς πόρους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε αυτόν τον τομέα σε ποιο βαθμό η παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο. Και σίγουρα εμείς θα καταθέσουμε και κάποιες τροπολογίες υποστηρίζοντας πιστεύω αυτά τα οποία είπε ήδη ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάντσε Σμιτ, το λόγο παρακαλώ. Συγγνώμη, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το κείμενο το οποίο να θέλετε πηγαίνει προς την κατεύθυνση που, των προτάσεών μου στην Επιτροπή Πολιτισμού. Είναι διτός ο χαρακτήρας Συμβάλλει επίσης στην κοινωνική ένταξη, στην κοινωνική ενσωμάτωση, στην διάδοση, αν θέλετε, την εξάπλωση της, της ευρωπαϊκής ταυτότητος που θα μπορούσε αν θέλετε, αν θέλετε να, ρίξει αν θέλετε τα φράγματα αν θέλετε, τα νοητικά. Συμβάλλει επίσης την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα των εδαφών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε επίσης και ο ψηφιακό τομέας διότι δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, δημιουργούν πλούτο και νομίζω ότι όλοι έχουμε επίγνωση πλέον του ρόλου, του σημαντικού ρόλου που μπορεί να παίξει, αν θέλετε, η πολιτική συνοχή στον τομέα αυτό. Που θα πρέπει βεβαίω να αξιοποιηθεί. Και αυτό αναφέρεται νομίζω πολύ σωστά στην έκθεση αυτή. Και το ρόλο δηλαδή μπορούν να παίξουν οι τοπικέ αρχέ στην προώθηση, στην προαγωγή, αν θέλετε, αυτών των πόρων θέλετε, συνοχή όπως επίσης και να συμπεριλάβουν δηλαδή στην πολιτική ανάπτυξη της περιφερειακής και της τοπικής αυτές αν θέλετε τις, τους κλάδους αν θέλετε, την δημιουργική δηλαδή και την πολιτιστική βιομηχανία. Αναφέρεται επίσης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η πρόσβαση στα διαστοτικά κονδύλια αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον τομέα όμως του πολιτισμού δηλαδή και της ε, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα μικρό επιτυχίε στην πρόσβαση στα κονδύλια αυτά. Αυτέ είναι οι παρατηρήσει που θέλω να κάνω. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πέτρη Ζήμαν έχει το λόγο τώρα. Yeah, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βλασάκ για την πλήρη αυτή έκθεση. Μία μικρή πρόταση για προσθήκη, αν συμφωνεί ο εισηγητής. Όταν μιλάμε για τον δημιουργικό τομέα, η κουλτούρα είναι ένα τμήμα αυτού του δημιουργικού τομέα, αλλά η δημιουργία ξεπερνάει τον στενό τομέα της κουλτούρας. Επίσης αναφέρεται στις ε, αδυναμίες που έχει αυτός ο τομέας ο κύριος Βλάσεκ. Θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία φορέων οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετούν και την κατάρτιση στους ε, δημιουργικούς τομείς και οι οποίοι συνδέουν τη δημιουργία με τι επαγγελματικέ δραστηριότητες. Υπάρχουν τέτοια κέντρα που προωθούν τη δημιουργικότητα σε, σε πολλές χώρες της Ευρώπης που δεν περιλαμβάνουν μονάχα την κουλτούρα αλλά πράγματα όπως η σχεδίαση για το ίντερνετ και άλλες δραστηριότητες πιο πρακτικές πολλές φορές. Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι φορείς οι οποίε ε, παίζουν σημαντικό ρόλο όπω και τα λεγόμενα κέντρα startup που παίζουν σημαντικό ρόλο. Επομένω, ίσω θα πρέπει να μην περιοριστούμε μονάχα στον πολιτιστικό τομέα, αλλά γενικά στον τομέα τη δημιουργία, ο οποίο στη Γερμανία είναι τόσο διαδεδομένο όσο και ο τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία Ευχαριστώ. Ο Μικαέλ Τόερερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Από την πλευρά των φιλελευθέρων θέλω και εγώ να κάνω μερικέ παρατηρήσει. Αναφέρθηκε η πράσινη βίβλος ήδη με την έννοια της ε, οικονομίας, της κουλτούρας και της δημιουργίας. Υπάρχουν και οικονομικά στοιχεία λοιπόν εδώ, για τα οποία θα ήθελα εγώ να τονίσω ότι οι πολιτιστικοί φορείς σε όλη την Ευρώπη παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και για, για την ε, διατήρηση της ε, πολυμορφίας και εφόσον βρισκόμαστε μέσα στο έτος της, του εθελοντισμού και εκεί μπορεί να υπάρξει ένας σημαντικός ρόλος. Μπορεί να είναι αντικείμενο διαμάχης τι είναι η κουλτούρα, πού σταματάει ο πολιτισμός, πού είναι τα όρια και επίσης το αν μπορεί να διατηρηθεί ο πολιτισμό χωρί δημόσιε επιδοτήσει. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, απλώ θέλω να υποστηρίξω την Κομισιόν σε αυτά που έκανε για το γεγονό ότι έθεσε στο κέντρο τη ε, προσοχή τη τον τομέα το δημιουργικό, τον τομέα τη κουλτούρα και εδώ θέλω να. Είναι καλό να δούμε ποιο είναι ο ρόλος και των επιδοτήσεων τη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και στόχοι δημόσιοι το να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια υποστήριξη της ε, χρηματοδότησης του τομέα αυτού και την άρση των εμποδίων που εμποδίσουν την, ε, ε, την πολιτιστική δημιουργία. Υπάρχουν και τα λεγόμενα προγράμματα φάρη τα οποία δεν αναφέρθηκαν από τον κύριο Σίμων, αλλά έχουμε παραγωγή χάρη προγράμματα όπως αυτό της Ακαδημίας του Μανχάιμ και αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να παίξει ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη. Για όλα αυτά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αναφερθούν όλα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι πρόκειται για περιορισμένες επιδοτήσεις το χρόνο, ότι πρόκειται κυρίως για χρηματοδότηση εκκίνησης για να περάσει ένας φορέας στο χώρο της αγοράς. Επομένως δεν πρέπει να μιλάμε μονάχα για αυτούς οι οποίοι παίρνουν μόνιμες επιδοτήσεις, αλλά κυρίως για την ενθάρρυνση της εκκίνησης. Επομένως είναι σημαντικό, όπως λέει και η Πράσινη Βίβλος, να τονίσουμε αυτή την πτυχή της χρηματοδότησης για εκκίνηση. Ευχαριστώ. Ο Θέλει να προσθέσει κάτι. Δεν επιμένω. Άμα θέλεις. Ε, ναι, Πρόεδρε. Πήρα πάρα πολλέ σημειώσει και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Η προθεσμένη διάθεση τροπολογιών είναι 3η Φεβρουαρίου, 6 το απόγευμα. Και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το σημείο 5. Έκθεση τη Σοφή Οκονή, μια νέα αγορά για τι επιχειρήσει και την ανάπτυξη. Σοφή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, που σας ε, προτείνεται εδώ και που στοχεύει την Επιτροπή ΙΜΚΟ, η οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας στο πλαίσιο λοιπόν της Επιτροπής ΙΜΚΟ τρεις εκθέσεις πρόκειται να καταπιστούν. Μία έκθεση για την ενιαία αγορά των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη, μία άλλη έκθεση για μια ενιαία αγορά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και μία τρίτη έκθεση για την διακυβέρνηση και την ε, σύμπραξη στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Σε αυτή τη γνωμοδότηση, Πρόεδρε, αλλά αυτή η γνωμοδότηση ήταν ουσιαστική σημασία για μένα, δηλαδή να υπάρξει συμμετοχή και παρέμβαση της πολιτικής συνοχής σε σχέση με την πράξη της ενιαίας αγοράς. Η ενιαία αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Η κοινή αγορά το 57 ενιαία αγορά σήμερα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει ένα βήμα περαιτέρω προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς προς όφελος των πολιτών αφενός αλλά και των επιχειρήσεων αφετέρου. Η σχέση ανάμεσα στην ενιαία αγορά και την περιφερειακή ανάπτυξη είναι πολύ στενή. Χρειάζεται λοιπόν η Επιτροπή μας να ε, συντάξει μια γνωμοδότηση για την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ σε θέματα που αφορούν την ενιαία αγορά. Θεωρώ πως η περιφερειακή πολιτική και η ενιαία αγορά είναι δύο πολιτικές άρρηκτα συνδεδεμένες και συρωματικές συνάμα και συμβάλλουν στην δημιουργία μιας Ευρώπης πιο ισχυρής γιατί έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Σε σχέση λοιπόν με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης να πω ότι χρειάζεται να συμπεριλάβει κάποιες δεσμεύσεις ε, πρώτα απ' όλα σε σχέση με τις τρεις εκθέσεις ε, της Επιτροπής ΙΜΚΟ εμείς ε, ως Επιτροπή ΡΕΖΙ μπορούμε να παρεύουμε μόνο στο πλαίσιο μιας μόνο γνωμοδότησης. Εμείς προτιμήσαμε λοιπόν την ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε πως αυτό είναι το επίκεντρο και το δυνατό στοιχείο της περιφερειακής πολιτικής και θα παρεύουμε λιγότερο για την διακυβέρνηση και την ελευθερική αγορά για την ε, ανταγωνιστικότητα. Τώρα για τις αυτές νομοδοτήσεις ε, γνωρίζετε ότι είμαστε πολύ περιορισμένοι σε ό,τι αφορά την ε, έκταση της νομοδότησης ε, σε σχέση λοιπόν με αυτή την νομοδότηση, εγώ επικεντρώθηκα στο εξή. Πρώτον, ότι ενέκρινα συνολικά το διάβημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνέδε την Επιτροπή Ρέζη σε αυτό το ζήτημα που άπτεται της, ενίας, της πράξης για την ενία αγορά για μας, για μένα ιδιαίτερα, δείχνει την δίνει την ευκαιρία για να ενισχύσουμε αυτή την ιδέα της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της, ε, ε, της Επιτροπής ε, Ρέζι. Και δεύτερον, θέλω να επενθυμίσω το ρόλο της περιφερειακής πολιτικής, όπως προείπα, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, ειδικά με την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών. Αυτό τι σημαίνει, ότι οποιοδήποτε και αν είναι ο τόπο εγκατάσταση μια επιχειρήση, ε, κατά το μάλλον ήταν απομακρυσμένο, ε, χρειάζεται η επιχείρηση αυτή να έχει μια ισότιμη πρόσβαση στο σύνολο τη αγορά. Και αυτή είναι η δύναμη ισχύ τη περιφερειακή πολιτική. Δηλαδή θα υπάρχει συνάμα μια εδαφική συνοχή αλλά και μια ε, και μια περιφερειακή συνοχή. Κάτι το οποίο ανάγγειλε και ο, ανήγγειλε και ο Επίτροπος Χάν στην έκθεση και κάτι ακόμα, στήριξη στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού που αφορά στην ε, περιφερειακή πολιτική. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτά τα ορατά αλλά και αόρατα σύνορα μέσα ακριβώς αυτή τη συνεργασία της εδαφικής. Και τρίτον, προτείνουμε κάποιες λύσεις και θα είμαστε συντονισμένοι με την ενία πράξη. Μπορείτε να διαβάσετε κάποιες λεπτομέρειες. Ε, θα σας αναφέρω μερικές από αυτές για να μην καταγραφτώ του χρόνου σας. Πρώτα απ' όλα η χρηματοδότηση καινοτόμων προγραμμάτων, μιλάμε για τα project bond, γιατί να μην έχουμε ε, δηλαδή, δυνατότητα χρηματοδότησης συγκεκριμένων σχεδίων ε, μέσω ομολόγων, ε, γιατί να μην μπορούμε να προσπαθήσουμε να πάμε παραπέρα, δηλαδή π.χ. τομέας μεταφορών. Παράδειγμα, μια δράση πιο αποφασιστική σε θέματα μεταφοράς των οδηγιών είναι επιτακτικό. Τα κράτη να εφαρμόσουν τις επιμέρους οδηγίες ε, και χρειάζεται να δείξουμε αποφασιστικότητα αναφορικά με τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Και επίσης ε, την ε, αύξηση του προπολισμού για θέματα εδαφικής συνεργασίας. Με τη Σνάλφο έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία. Η περιφερειακή αυτή η εδαφική αυτή συνεργασία είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και θεωρώ ότι πρόκειται για στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε εντελεχέστερα από κοινού. Τώρα για την νομοδότηση έχουμε ένα timing, κάποιος ε, προγραμματισμό χρονικό, ένα χρονισμό και εσείς κυρία Πρόεδρε θα μας πείτε τις ρίες. Η έγκριση στην Επιτροπή Ρέζουση θα πρέπει να γίνει στις 23 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δύο ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια στην Επιτροπή αυτή και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, είναι πολύ καλές οι προτάσεις της και εξάλλου υπάρχουν κάποια σημεία που θεωρώ ότι η Περιφερειακή Επιτροπή έχει ιδιαίτερη ευθύνη και αρμοδιότητα στα σημεία αυτά και εκεί θα πρέπει εμεί να εστιάσουμε την προσοχή μας και να καταθέσουμε τροπολογίες. Θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια, παραδείγματο χάρη, να αντιμετωπίσει το θέμα των δημοσίων προμηθειών. Η εισηγήτρια είπε ότι θα πρέπει εδώ να υπάρξει και μια αξιολόγηση και αυτό ε, αναφέρθηκε και στην έκθεση του συναδέλφου για τις δημόσιες προμήθειες. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να υπάρξει για κάποια διατύπωση που να λέει ότι η Επιτροπή μας περιμένει ότι αυτές οι δημόσιες διαδικασίες διαγωνισμού θα μπορούν να διέπονται από μεγαλύτερη ευφελιξία και επίσης να έχουν και μια μεγαλύτερη απλοποίηση. Είναι ένα σημείο ο κύριος Φλάσεκ, συγγνώμη, ξέχασα το όνομά σας, ο κύριος Φλάσεκ προφανώς έχει γράψει την έκθεση, συγγνώμη που δεν μου ήρθε στο νου το όνομά σας. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί στην έκθεση για να κατανοήσει η Κομισιόν ότι είναι απαραίτητο να προβλέψει και μία αξιολόγηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να το αναφέρουμε. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να δω να αντανακλάται σε αυτή την έκθεση είναι το θέμα της συνεργασίας. Η συνθήκη της Λισαβόνας ζητάει σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό να υπάρξει συμμετοχή σε όλες αυτές τις ενέργειες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στις, επίσης στο εγγραφό της στις διαβουλεύσεις με τους Δήμους και τις κοινότητες. Και εγώ βρίσκω ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι βάσει των παραδόσεων στι περιοχέ αυτέ θα πρέπει να συμμετέχουν τοπικέ αρχέ, συνδικάτα κτλ. Ενώσει. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο το οποίο λέει η πρόταση τη Κομισιόν. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να ενισχύσουμε ιδιαίτερα την συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και επίσης να τονίσουμε και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής των Περιφερειών γιατί οι κοινότητες και οι δήμοι είναι αυτοί που σε τελική ανάλυση εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, επομένως θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μπορούν να έχουν και κάποια συμμετοχή στη διαμόρφωση <clears throat> του ευρωπαϊκού δικαίου. Επίσης το ζήτημα του πακέτου για την παροχή ε, υπηρεσιών στην περίπτωση αυτή των ε, δημοκή και επίσης θέλω να αναφερθώ και στο σύστημα ΙΜΗ, e το οποίο παρουσιάζεται από την Κομισιόν ως ένα καλό υπόδειγμα για την ευρωπαϊκοποίηση των Δήμων και Κοινοτήτων. Αλλά κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο σύστημα. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε προηγουμένως να το αξιολογήσουμε και να δούμε πώς απέδωσε προτού θελήσουμε να το μεταλαμαδεύσουμε σε άλλες περιοχές, σε άλλους χώρους. Τέσσερις εισηγητές έχουμε. Η κυρία Βέσφαρ. Ξεκινώ με κάποιες ε, γενικές παρατηρήσεις στα θέματα αυτά. Το κείμενο για την έννοια αγορά ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Δυστυχώς, αν δούμε το μεταγενέστερο κείμενο της Κομισιόν, δεν υπάρχει μια πολιτική ιδέα για να μπορέσει να προωθηθεί περισσότερο αυτή η ιδέα ακόμα και αν είναι απαραίτητο να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει ένας συνδετικός ιστός που να συνδέει τα διάφορα τα οποία προτείνει η Κομισιόν, τα οποία είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος ονίων, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα μέτρα για την υλοποίησή τους. Το πακέτο της Κομισιόν ξεκινάει έχοντας υπόψη το επιχειρήν και μόνο μετά περνάει στους καταναλωτές. Αυτό δείχνει ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι η καρδιά της εσωτερικής αγοράς δεν είναι οι πολίτες, αλλά οι επιχειρήσεις. Ίσως η Κομισιόν δεν έχει να μας προσθέσει καμία ιδέα για τις λεγόμενες αξιολογήσεις σε κοινωνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα μέτρα της εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι για τη γενική έκθεση και τώρα στέκομαι στην γνωμοδότηση. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Οκονή, η οποία είναι η συντάκτρια της γνωμοδότησης. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το σχέδιο γνωμοδότησής της και παρέχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις που έχουν την υπογραφή, έχουν το ύφο της Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε κάποιες, ε, ε, κάποια αιτήματα τα οποία θα τα παρουσιάσουμε υπό τη μορφή τροπολογιών και θα αναφέρω κάποια από αυτά. Καταρχήν, στο σημείο 1 της γνωμοδότησης, εμείς χαιρετίζουμε τις προτάσεις της Κομισιόν γενικά και εμείς. Αλλά είπα ότι δεν είναι επαρκής ήδη. Αλλά ιδίω εμείς λυπούμεθα ότι το, το, η πρόταση της Κομισιόν δεν προβλέπει καθόλου το να υπάρξει μια ρήτρα για την αξιολόγηση σε κοινωνικό επίπεδο των μέτρων αυτών. Στο σημείο 4 της ε, γνωμοδότησης προκύπτει το γεγονός ότι είναι σημαντική αυτή η διαδικασία για τις περιφέρειες, αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι και οι περιοχές, οι περιφέρειες της Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντικές για, ε, ε, την περιφερειακή πολιτική. Είναι αμφίδρομη λοιπόν η σχέση των, των δύο. Είναι επομένω απαράγραπτη μια σωστή περιφερειακή πολιτική για την περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης. Θα πρέπει να τονιστεί λοιπόν ιδιαίτερα ποια είναι η σημασία που επέχουν οι περιφέρειες και η ανάπτυξή τους για την εσωτερική αγορά. Στο σημείο 7 αναφέρεται η αρχή της εξάρτησης και εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει κανείς να αναφέρει όπως σωστά έπραξε και η κυρία Οκόνη για μένα υπάρχει το ερώτημα του αν αυτή η αρχή της ε, της εξάρτησης της, ε, των προϋποθέσεων μπορεί να τύχει χρήσεων επίσης. Αυτή η, η προβληματική δεν ξέρω αν είναι ένα θέμα το οποίο εμείς θα πρέπει να το αναλύσουμε περισσότερο στην ε, γνωμοδότηση. Μέσα σε ένα σύντομο πάντως χρονικό διάστημα πρέπει να τονίσω ότι η κυρία Κονή κατάφερε να συντάξει μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. κύριος Βλασέκ. Ο κύριος Βλασέκ. Ευχαριστώ. Θέλω να τονίσω την θετική μου στάση εναντί αυτής της έκθεσης. tady se shoduji s paní Ríle, že je nemůžeme nějakým způsobem vinout. you speak a beautiful language, but we don't have translation, I think. No, okay. at least I don't have. I... I would like to stress that the role of uh, local and regional municipalities is also very strong. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Από την άλλη και αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται. Να πω επίσης θα ήθελα ότι από πρακτική σκοπιάς γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει οι τουριστικές περιοχές. Οι υποδομές δηλαδή οι οποίες δεν είναι οι κατάλληλες και θα πρέπει να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας του περιβάλλοντος δηλαδή και νέων υποδομών. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αγκουράκης τώρα έχει το λόγο παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι αν ήταν να προσφέρουμε ουσιαστική υπηρεσία στις συζητήσεις και τις εξελίξεις έπρεπε η έκθεσή μας να απορρίψει την ε, ενιαία αγορά και να πει ότι όσον αφορά ε, τα αποτελέσματά της είναι καταστροφικά. Συζητάμε, κυρία Πρόεδρε, σε μια εποχή που έχουμε 20 εκατομμύρια ανέργους, που τίθεται υπό αμφισβήτηση αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει, συζητάμε σε μια εποχή που μιλάμε για μηχανισμό στήριξης, ε, ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και ακόμα θέλουμε να βαθύνει ακόμα περισσότερο η ενιαία αγορά συζητάμε για μια εποχή, κυρία Πρόεδρε, όπου οι περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της ενιαίας αγοράς και θα έπρεπε ως Επιτροπή Περιφερειών να εστιάσουμε σε αυτό το ζήτημα και δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Έχουμε μια έκθεση, λες και είμαστε στο πρώτο χρόνο της ενιαίας αγοράς, λες και δεν, δεν υπάρχουν δεκάδες μέτρα τα οποία ακριβώς αυτό θέλουν. Την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και μας, δεν, μας, δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτό το ζήτημα. Συγγνώμη που μιλάω έτσι κυρία Πρόεδρε, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο όπου η Ουγγρική Προεδρία ζητάει σπόνσορες για να εκδώσει το πρόγραμμά της και έχουμε την Volkswagen, τη Siemens, την ε, Samsung στο εξώφυλλο της Ουγγρικής Προεδρίας και εμείς μιλάμε για την νέα αγορά που θα μας πάει μπροστά. Νομίζω ότι ειδικά οι περιφέρειες υποφέρουν από αυτή την υπόθεση και όπως πολύ συχνά έχουμε πει σε αυτή την ε, αίθουσα τα προγράμματα συνοχής ε, ε, ήρθαν για να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ενιαίας αγοράς. Κατά συνέπεια νομίζω θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο κριτικοί και να απορρίψουμε την έννοια της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Η κυρία Σάντζου Σμιτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχήν να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για το περιεχόμενο τη γνωμοδοτήσεώ του. διότι αξιοποιεί την εδαφική ή την περιφερειακή συνεργασία όσον αφορά την εμβάθυνση τη εσωτερική αγορά, τη ενιαία αγορά. Οι παραμεθόριε ζώνε είναι ζώνε, αν θέλετε, που παρουσιάζουν, αν θέλετε, ελλείψει ανταγωνιστικότητα για τι επιχειρήσει, λόγω, αν θέλετε, των διοικητικών, αν θέλετε, κανονιστικών εμποδίων. Και, αν θέλετε, τι διαφορετικέ ενισχύσει που δίνουν τα κράτη-μέλη στι περιφέρειε. Η διασυνορική συνεργασία, συνεπώ, αποτελεί, αν θέλετε, ένα πραγματικό ορυχείο ανάπτυξη που πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσουμε τα σύνορα είναι ένα τόπο αν θέλετε, εμβάθυνση τη ενιαία εσωτερική αγορά, Αν η εδαφική συνεργασία, ε, αν θέλετε, μειώνει αν θέλετε, τα προβλήματα αυτά, ειδικότερα για του πολίτε. λέτε ότι οι πολιτε πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο τη εσωτερική αγορά και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, αν θέλετε, τη περιφερειακή πολιτική. Προφανώ λοιπόν, τάσσομαι υπέρ τη ενίσχυση του προπολογισμού τη εδαφική και περιφερειακή συνεργασία. Αυτή η γνωμοδότηση μου δίνει, αν θέλετε, ένα επιπλέον επιχείρημα επίσης ότι είναι ε, μια πολιτική επενδύσεων και όχι παροχής βοήθειας. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι δεν εξυπηρετεί και που στρεβλώνει δηλαδή την, ε, τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορών οικονομικών φορέων και παραγόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανής Λερόι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό το ότι αντιδρούμε για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση και την περάτωση της εσωτερικής αγοράς. Αναφέρθηκε η εδαφική διάσταση, η οποία είναι πολύ σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχυθεί η εδαφική αυτή συνοχή και να έχουμε μια καλύτερη διατύπωση αυτών των εργαλείων. Εδώ μιλάμε περισσότερο για δραστηριότητες που έχουν διαμεθοριακό χαρακτήρα και πρέπει να είναι σαφές ότι θα πρέπει οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίζουν επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ένθεν και εκείθεν των συνόρων. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλες τις ενδιάμεσες κατηγορίες οι οποίες πολλές φορές δεν κατατάσσονται εύκολα σε μία ή άλλη κατηγορία. Όλα αυτά έχουν σαν στόχο την καλύτερη ανταγωνιστικότητα και την σύγκληση. Ίσως θα πρέπει να δοθούν και ενδιάμεσες ε, να και ενδιάμεσες λύσεις, αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την ε, κατεύθυνση αυτή η οποία διαγράφεται στη γνωμοδότηση αυτή. Εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη όλο και περισσότερο περνάει σε μία η δίκευση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε περιφέρεια της Ευρώπης ειδικεύεται περισσότερο. Μία παράγει αυτοκίνητα, μία έχει βιοτεχνολογία κτλ. Όλα αυτά θα έπρεπε να μας οδηγήσουν να σκεφτούμε καλύτερα για μία μορφή δημιουργίας συμπλεγμάτων, clusters για τις δραστηριότητες. Έχουμε μία διαδικασία η οποία οδηγεί στην ε, μεγαλύτερη ειδίκευση και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Πρέπει λοιπόν οι επιδοτήσεις να έχουν σαν στόχο να επιτύχουν καλύτερη ενσωμάτωση. Παραδείγματο χάρη στην Ελλάδα να υπάρχει χρήση των περιφερειακών πόρων για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιφερειών στην εσωτερική αγορά. Δεν πρέπει να λέμε ότι οι περιοχές αποκλίνουν. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε την ε, σύγκλησή τους χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά και τα περιφερειακά μας εργαλεία ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανασύγκλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την γνωμοδότηση της συναδέλφου Οκονή ε, η οποία νομίζω δίνει τις ε, πολύ σωστές ε, συστάσεις στην αρμόδια της επιτροπή. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας οδηγεί στο να αναρωθούμε σε μια σειρά, για μια σειρά θεμάτων για τα οποία η Επιτροπή θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, ειδικά σε ό,τι αφορά την μελλοντική ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής αλλά και της πολιτικής συνοχής. Χαίρομαι που μπορώ να συμφωνήσω και με τις προτάσεις ορισμένων ε, σκιωδών εισηγητών πως ε, αυτό το ζήτημα θα πρέπει να ε, ξεκινάει από τον πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να είναι το επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς, της ενίας αγοράς. Εμείς αυτό είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και στην Επιτροπή της οποίας προεδρεύει και έχουμε συντάξει μια γνωμοδότηση. Αναφέρομαι στην Επιτροπή Αναφορών που στόχος μας είναι η προστασία των πολιτών και επικεντρώσαμε την προσοχή μας στο ζήτημα της ιδιαίτερης προστασίας που θα πρέπει να μας απασχολήσει για την προστασία των καταναλωτών. Αυτό το θέμα δεν θίγεται στη γνωμοδότηση. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των της ε, Περιφερειακής ε, Επιτροπής σε συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών για την πρόθεση μιας πολιτικής συνοχής, μια περιφερειακή συνοχή, η οποία έχει ως στόχο την υπέρβαση των ανισοτήτων και ανισορροπιών προκειμένου να δημιουργήσει συνθήκες ισότητας για όλους. Συμφωνώ στο σημείο 7 με το ερεσιμότητα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να μας απασχολήσει αλλά καλό να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν εισάγουμε αυτό το θέμα διότι όπως πολύ σωστά και η συνάδελφος Οκονή την γνωμοδότησή της πρέπει να ε, τύχει κάποια κατεύθυνση και καθοδήγησης και να μην αφαιθεί ελεύθερο σε ένα πλαίσιο των συζητήσεων. Και τέλος, ε, η περιφερειακή πολιτική είναι μια πολιτική επενδύσεων αλλά και ανάπτυξης. Και ανάπτυξη, κατά την άποψή μου, δεν σημαίνει μια ε, πολιτική πρόνοιας, αλλά θα πρέπει να την υπόψη οι διαφορές οικονομικές, κοινωνικές που υπάρχουν ανάμεσα στις περιοχές προκειμένου να τις υπερβούμε. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χορηγούμε μόνο βοήθεια και επιδοτήσεις, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις περιφέρειες. Ευχαριστώ. Thank you very much. please. Ο κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν ήθελα καταρχήν να λάβω το λόγο, αλλά με εν τη συζητήσεως έχει έρθει στο πνεύμα μου το ότι είναι σημαντικό να τονίσω ότι στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης μαζί με την έκθεση αυτή να κάνουμε κάποια διευκρίνηση ορισμένων θέσεων ή να κάνουμε ένα καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ διαφορετικών ενίων. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε σωστά, αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Είναι σαφές ότι η περιφερειακή ε, πολιτική έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει και ανισομέρειες οι οποίες δημιουργούνται στον οικονομικό τομέα μεταξύ κρατών μελών ή και μέσα στα κράτη-μέλη. Εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες υπολείπονται ε, οικονομικά σε περιοχές όπου υπάρχει και υστέρηση στον πολιτιστικό τομέα, σε τομέα συμμετοχή στην ε, γενικότερη οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι σε μια προοπτική όπου βλέπουμε να αυξάνεται ο παγκοσμίος πληθυσμός και να μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι, εμείς θα πρέπει να αυξήσουμε μεν την ευμάρεια και την, ε, στο επίπεδο της ευρωπαϊκής έννοιας, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μείωση των ε, ανισομεριών χωρίς να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να απομακρυνθούμε από την αγορά. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά αυτά τα οποία ε, ανέφερε ο συνάδελφος ε, Γκουράκη σε σχέση με το ρόλο της αγοράς. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε μια λαθασμένη κατεύθυνση ή να έχουμε μια λαθασμένη εντύπωση. Δείχνουν τα στοιχεία τα αριθμητικά ότι η εσωτερική αγορά και η εισαγωγή τη εσωτερική αγορά οδήγησαν σε μια αύξηση τη ευμάρεια σε όλη την Ευρώπη παρά το γεγονό ότι μπορεί να υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες. Ορισμένες κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα ενώ άλλε δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν αυτά τα πλεονεκτήματα και αυτό δεν αφορά ορισμένες μονάχα χώρες, ακόμα και στις ισχυρότερες οικονομίες εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν τα έχουν καταφέρει τόσο καλά. Επομένως, τίθεται το θέμα του ποιος πρέπει να είναι ο στόχος της περιφερειακής πολιτικής και τώρα είμαι ευγνώμων στο γεγονός, για το, για, στην εισηγήτρια για το γεγονός ότι έχει ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση η εισηγήτρια σε σχέση με τον ρόλο της Περιφερειακής Επιτροπής. Αυτά τα τόνισε και η κυρία Ματσόνη. Είπαμε ότι πρέπει ουσιαστικά να δώσουμε βοήθεια για αυτοβοήθεια στις ε, περιφέρειες, να μπορέσουν να δημιουργήσουν υποδομές, να δημιουργήσουν δομές ε, που θα προσελκύσουν επενδύσεις, θα βοηθήσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επομένως, η περιφερειακή πολιτική έχει σαν αποτέλεσμα να βοηθήσει τις περιοχές να, να έχουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και αν αυτό γίνει κτήμα όλων μας, θα καταλάβουμε ότι με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται και οι στόχοι της εσωτερικής αγοράς. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τον Μάριο Μόντι, με τον Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά, να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα και τα θέματα τα οποία έχουμε εμείς αναφέρει με κάποιο κριτικό πνεύμα από την Επιτροπή ε, Περιφερειακής Επιτροπής, να μπορέσουμε να τα αντιπαραθέσουμε με την άποψη της Κομισιόν. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τη συζήτηση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ λέει και η πρόεδρο. Ο Φρανσουά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα έκθεση και φαίνεται από το γεγονός ότι πολλοί έλαβαν το λόγο για το θέμα αυτό. Είναι ένας χώρος Δυναμικότητα που δημιουργεί μεγαλύτερη δυναμική για τι οικονομίες η ενιαία αγορά και επομένω δίνει περισσότερε δυνατότητε για το επίπεδο το βιωτικό των πολιτών τη Ευρώπη, αλλά εκφύσεω η εσωτερική αγορά δεν περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία εξισορρόψη και ισορροπία που είναι απαραίτητα για όλε τι κοινωνίε. Η Κομισιόν στην πρότασή τη εξάλλου μιλάει στην έκθεσή της για την ενίσχυση τη αλληλεγγύη. στην εσωτερική αγορά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχει, ένα πρόβλημα το οποίο έχει η ενή αγορά από τα γενοφάσκα της. Δεν είναι κάτι το οποίο όταν το λέω αυτό είναι μια ιδεολογική δίκη προθέσεων. Ο στόχος είναι να υπάρξει ισορροπία, αλλά ξέρουμε ότι η εσωτερική αγορά βοηθάει τις πλούσιες περιοχές περισσότερο από τις μειονεκτικές περιοχές. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα αντιστάθμισμα, μια ρύθμιση για τα θέματα αυτά. Και αυτό είναι ένα ασθενικό, ένα ασθενές σημείο στην έκθεση της Κομισιόν <clears throat> ότι μεταξύ των 56 προτάσεων που αναφέρει δεν υπάρχει τίποτα σε σχέση με την ανάγκη να υπάρξει επάνεξη και ίσως η εισηγήτρια μπορεί να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Οκονή, θέλετε να κάνετε κάποια καταληκτικά σχόλια ή όχι. Να πω ότι Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, όλες τις παρεμβάσεις και τα σχόλια. Θα τα λάβω υπόψη μου και για να διαφωνήσω τον Λάμπερτ Βανιστερόε να του πω ότι σε ό,τι φορά τις ενδιάμεσες κατηγορίες εγκύψατε επί του ζητήματος για να δείτε πώς ε, αν οι περιφέρειες που δεν μπορούν παρά να βασιστούν στο phasing out παρά μόνο μία φορά στον προγραμματισμό, το ενδιάμεσο σύστημα δεν νομίζω ότι είναι πιο σίγουρο και πιο ασφαλές και ότι θα μπορούσε να ενισχύσει το σύνολο της πολιτικής συνοχής. Αυτή είναι η εντύπωσή μου σε σχέση με αυτό το άρθρο 6 της ενδιάμεσης κατηγορίας. Ευχαριστώ. Ολοκλώσαμε την συζήτηση επί της νομοδοτήσεως. Να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την τροπολογιών είναι η 7η Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα και επίσης δύο ακόμα εκθέσεις που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή η έκθεση του κυρίου Γκάιερ για την επαλλαγή 2009 και του κυρίου Καρόνα ε, σχετικά με την Ευρώπη ως πρώτο τουριστικό προορισμό και σε συμφωνία με τους εισηγητές θα προσπαθήσουμε να τις περιλάβουμε στο αυριανό μας πρόγραμμα. Τώρα έχουμε την συνάντηση με την Ουγγρική Προεδρία. Ο Υπουργός ε, ήδη βρίσκεται ανάμεσά μας. Ως εκ τούτου μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 9 της Διατάξεως. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να λάβετε τις θέσεις σας, γιατί ξεκινάει η συνάντηση και πάλι. Έχουμε ανάμεσά μας, μαζί μας, τον Υπουργό Τόμας Φελέτζε, της Ουγγρικής Κυβερνήσεως επακεφαλής του Υπουργείου Εθνικής Ανάπτυξης, καθήκοντα του οποίου είναι και η πολιτική συνοχής κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής ο Υπουργό εργάζεται εδώ στι Βρυξέλλε. Έχει συνεδρίαση μετά από συνεδρίαση. Είχε μάλλον σήμερα. Ελπίζω να επιβιώσετε μετά τη σημερινή σα συνάντηση μαζί μα. Αλλά ε, θέλουμε να σα ακούσουμε και θέλουμε πολύ καλέ σχέσει μαζί σα κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα. Θα ξεκινήσουμε με τα εισαγωγικά σχόλια του Υπουργού, αγαπητοί συνάδελφοι, και κατόπιν θα ξεκινήσουμε μια ανταλλαγή απόψεων ή την υποβολή ερωτήσεων από πλευρά σα. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλου σα να καθίσετε για να μπορέσουν να ξεκινήσει αυτή η συνάντηση. Όσοι από εσά έχετε και θέλετε να έχετε άλλε συζητήσει, παρακαλώ να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Ξεκινήσατε. Okay. Uh, thank you very much, uh, Madam Chairperson. Uh, I hope everybody hears me. Ελπίζω να με ακούτε όλοι σας. Προτού αλλάξω γλώσσα και να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας στα Ουγγρικά, θα ήθελα εν συντομία και εντάχει να σας συστηθώ και να σας εξηγήσω τις ευθύνες τις οποίες έχω αναλάβει στο Εθνικό Υπουργείο Ανάπτυξης της Ουγγαρίας προεπταμίνου δημιουργήθηκε αυτή η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Στην οποία υπάρχει και ένα σύστημα ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων. Δημιουργήθηκε ένα Υπουργείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Πόρων, Υπουργείο Εθνική Ανάπτυξη, το οποίο λαμβάνει υπόψη του και τι πολιτικέ ανάπτυξη τη χώρα στο σύνολό τη, την ενέργεια, το κλίμα δηλαδή, τι μεταφορέ, τι τηλεπικοινωνίε, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θέλετε, του κράτου και τη ε, πολιτική αν θέλετε κρατικών προμηθειών. Αυτό είναι το φάσμα θέλετε, των θεμάτων που απασχολούν το Υπουργείο μου. Και εντό του Υπουργείου αυτού έχω αναλάβει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να εκπροσωπώ την Ουγγρική κυβέρνηση στον τομέα τη πολιτική συνοχή και τη περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γυρίζω τώρα στα Ουγγρικά για να παρουσιάσω το πρόγραμμα τη Ουγγρική Προεδρία. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ουγγρική Προεδρία θέλει να παρουσιάσει το πρόγραμμά της για την συνοχή και φυσικά αυτό συνδέεται με μία σειρά από νομοθετικά μέτρα. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να προωθήσουμε ορισμένα μέτρα κλειδιά και να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να προωθήσουμε μια σειρά από εξελίξεις. Επίσης θέλουμε να φέρουμε στο τέλος του εξαμήνου μας τα θέματα της περιφερειακής πολιτικής στην, ε, στα χέρια της επερχόμενης Πολωνικής Προεδρίας με τέτοιο τρόπο ώστε το 2013 να έχουν περατωθεί μια σειρά από κέρια εγχειρήματα η περιφερειακή πολιτική πολλές φορές την χάνει συζήτηση κυρίως σε άτυπο επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών. Η Ουγγρική Προεδρία όμως θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πολιτική. Εγώ έχω την τιμή να εκπροσωπήσω λοιπόν την ε, Ουγγρική Προεδρία στις προσπάθειες αυτές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Εμείς γνωρίζουμε το έργο της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρουμε ότι εσείς έχετε μια στεναρή υποστήριξη υπέρ της περιφερειακής πολιτικής. Η θέση σας, η αντιμετώπιση σας για τα διάφορα προβλήματα είναι πάντα μια πηγή υποστήριξης για μας. Μας βοηθάτε για να έχουμε μια βελτίωση, μια ανάπτυξη των πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όσο και η Κομισιόν θα μπορέσουν να έχουν τη σωστή συνεργασία προς το κοινό συμφέρον. Και η Ουγγρική Προεδρία είναι έτοιμη να σας πληροφορήσει σε τακτά διαστήματα για την πρόοδο των εργασιών. Είναι πεπισμένη η Ουγγρική ε, Προεδρία ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η πολιτική περιφερειακών θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό θα προσδώσει και περαιτέρω αποτελεσματικότητα στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούνιο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν όλα αυτά τα θέματα να καταλήξουν στο Συμβούλιο Κορυφής του Ιουνίου. Η Ουγγρική Προεδρία έχει θέση στην ε, την περιφερειακή πολιτική και στην μέση διάταξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Εξάλλου θα υπάρξουν άτυπες συνεδριάσεις το Μάιο σε ό,τι αφορά τα θέματα της εδαφικής ανάπτυξης που θα λάβει χώρα στην Ουγγαρία, μια άτυπη σύνοδος υπουργών Χαιρετίζουμε και την πέμπτη έκθεση της Κομισιόν για τα θέματα συνοχής. Συμφωνούμε με τις προτάσεις και τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση αυτή και η πεποίθησή μας είναι ότι χρειάζονται ακόμα περισσότερες ενέργειες και περισσότερες διαπραγματεύσεις για να προωθηθεί περαιτέρω το θέμα αυτό. Θα αναφερθώ τώρα σε ορισμένα κέρια ζητήματα. Ε, εν ώψη των προηγουμένων εξελίξεων μπορώ να σας πω ότι όλα τα κράτη-μέλη θέλουν να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει μια στεναρή πολιτική συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Βέβαια, έχει καταστεί σαφές ότι χρειάζεται να, υπάρξει μια να υπάρξουν και κάποιες τροποποίησεις στην πορεία πλεύσεως, αλλά πάντα διατηρώντας την ενότητα της πολιτικής συνοχής, δίνοντας έμφαση στα αποτελέσματα και στην ενότητα αυτής της πολιτικής. Η πολιτική αυτή λοιπόν δεν πρέπει να δημιουργηθεί εκ του μηδενός, αλλά μπορεί να είναι αναγκαίο να υπάρξει μια νέα κατανομή πόρων, ώστε η κάθε, το κάθε κράτος μέλος να μπορεί να χρησιμοποιήσει με τον πιο επωφελή τρόπο αυτούς τους πόρους για να ενισχύσει την δραστηριότητα και την σύγκληση Επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί η περιφερειακή πολιτική και υπό το πρίσμα της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η οποία πρέπει να επιτευχθεί. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να έχουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε επίπεδο ε, υποδομών που θα αυξήσουν και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της οικονομικής κρίσης φυσικά είναι περιορισμένη οι πόροι στη διάθεσή μας και γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια αυτή η πόρη να χρησιμοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό και επωφελή τρόπο δυνατό. Θα πρέπει να μειωθούν οι περιτές ε, γραφειοκρατικές διαδικασίες και να απλοποιηθεί η διαδικασία για τη λειτουργία των περιφερειακών ταμείων. Δεν θέλουμε να θίξουμε την αυστηρότητα του ελέγχου, αλλά θέλουμε συγχρόνως να έχουμε μια καλύτερη λειτουργία και απλοποίηση των κανόνων, ώστε να μην υπάρχουν σφάλματα που προκύπτουν λόγω της πολυπλοκότητας των κανόνων. Επίσης, θέλουμε τα διάφορα νομοθετήματα τα οποία διέπουν τον τομέα αυτό να προσαρμοστούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα διάφορα ε, αιτήματα των κρατών μελών. Η Ουγγρική Προεδρία, εν προκειμένου, θα ασχοληθεί με τα εξή θέματα. Καταρχήν, οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 να εξυπηρετηθούν και να εστιάσουμε στα θέματα αυτά, να υπάρξει μια υποστήριξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης που συνάπτονται με το πρόγραμμα συνοχής. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα και συστήματα τα οποία θα προωθήσουν καλύτερη συνεργασία και συντονισμό και επίσης θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια καλύτερη ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής. Το πιο σημαντικό είναι η ενσωμάτωση στους στόχους της Ευρώπης 2020 και θέλουμε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στους στόχους κλειδιά της Ευρώπης 2020. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει μια μεγαλύτερη ενσωμάτωση και υποστήριξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τα δύο θα πρέπει να συμβαδίζουν απόλυτα. Πρέπει να σας πω επίσης ότι η πολιτική, η πολιτική συνοχής δεν είναι το μόνο εργαλείο της ε, στρατηγικής Ευρώπης 2020, αλλά συγχρόνως είναι και ένα εργαλείο το οποίο ενισχύει την εσωτερική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να μπορέσουν να συμβάλλουν ενεργά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παραμείνουν ισχυρά σε ανταγωνιστικό επίπεδο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μέλλον. Και έχουμε τώρα την λεγόμενη place-based αντιμετώπιση η οποία βασίζεται σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα απαράγραπτο εργαλείο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Νομίζουμε ότι ένα από τα καλύτερα επίπεδα, από τα καλύτερα παραδείγματα μάλλον, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης αφορά ακριβώς τη χρησιμοποίηση του τοπικού επίπεδου. Είναι πολύ σημαντική η στρατηγική για την Ευρώπη 2020, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πολυμορφία των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς μια πραγματική ισχυρή πολιτική συνοχή δεν μπορεί να υπάρξει μια ισχυρή Ευρώπη. Από τη μία πλευρά, επομένω πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε, στα κέρια θέματα και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των πολιτικών κατατομής και ότι θα εξασφαλιστεί και μια ισορροπία μεταξύ μιας ολοκληρωμένης αφενός πολιτικής και μεμονωμένων πολιτικών κατατομής. Η πολιτική συνοχή επίσης απαιτεί να υπάρξουν πολιτικές οι οποίες βασίζονται στην εμπειρογνωμοσύνη και οι οποίες είναι αξιόπιστες. Πρέπει να διέπεται από την αρχή της αλληλεγγύης και της ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης των διαφορετικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε περιφέρειες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν διαρθωτικά προβλήματα και εδώ εμπλέκεται προφανώς και το ενδιαφέρον των ιδίων των κρατών μελών. Είναι απαραίτητο να είναι ορατή και αποτελεσματική η πολιτική συνοχή, αλλά μα ενδιαφέρει επίση να είναι και μια ε, πολιτική εστραμμένη στα αποτελέσματα που θα αποδώσει συγκεκριμένου καρπού. Επιπλέον είναι απαραίτητο να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα καταμέτρηση τη απόδοση αυτών των πολιτικών. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε δείκτε οι οποίοι είναι διαφανεί και αξιόπιστοι και θα μπορέσουν ανεξάρτητα από άλλες οικονομικές διαδικασίες να μας καταδείξουν ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία προέρχονται από την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής. Αυτά φυσικά είναι και στοιχεία αξιοπιστίας αυτής της πολιτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά κυρίως σε τοπικό επίπεδο έτσι μονάχα μπορεί να επιτευχθεί μια μεγαλύτερη αποδοχή αυτών των πολιτικών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια σειρά από κίνητρα και εδώ η αιρεσιμότητα ως μηχανισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και η δυνατότητα ίσης πρόσβασης στα κοινωτικά κονδύλια είναι επίσης σημαντικό. Οποιαδήποτε κίνητρα δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μονάχα στην πολιτική συνοχή, αλλά και στα πλαίσια άλλων συναφών πολιτικών. Το σύστημα των αμοιβών και των κυρώσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο σόφρονα αλλά και επιφυλακτικό. Η πολιτική αυτή είναι ένα από τα καλύτερα και τα πιο σημαντικά εργαλεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι μια πολιτική η οποία υπερβαίνει τους απλούς τομείς και έχει μια γενικότερη στρατηγική αντιμετώπιση που είναι και εδαφική και αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ των περιοχών. Η πολιτική αυτή επίσης είναι μια πολιτική η οποία αναζητεί συνέργειες με άλλες πολιτικές. Η Ουγγρική Προεδρία ελπίζει ότι θα καταβληθούν όλες αυτές οι απαραίτητες προσπάθειες μέσα ώστε και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να υπάρξει κατάλληλη συνεργασία. Είμαστε πεπισμένοι ότι ιδίως λόγω της κρίσης είναι απαραίτητη η καλύτερη σύνδεση μεταξύ αυτών των πολιτικών. Οι περιοχές οι οποίες είναι υπολοιπόμενες, είναι μειονεκτικές, έχουν να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα προβλημάτων. Μπορούν να, το, να επιτύχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά μονάχα αν παραμείνει ε, το, η λειτουργία του κοινωνικού ταμείου στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Είναι απαραίτητο να προωθήσουμε και την διαφάνεια και την ορατότητα αυτής της πολιτικής κάτι το οποίο πρέπει να ισχύει και για την εφαρμογή του κοινωνικού ταμείου. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητη μια απλοποίηση σε πάρα πολλούς χώρους, το άχθος, το γραφειοκρατικό το οποίο συνοδεύει, πάρα πολλά προγράμματα θα πρέπει να μειωθεί. Πάντα μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανονισμού και πάντα μέσα στα πλαίσια ενός μοντέλου εποπτείας το οποίο έχει αναφερθεί και στην πέμπτη έκθεση συνοχής της, Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, είναι απαραίτητο να επιληθούν τα πλέγματα προβλημάτων τα οποία έχουν αναφερθεί και στην έκθεση της Κομισιόν. Είναι πολλά λοιπόν αυτά τα εγχειρήματα τα οποία είναι απαραίτητα στον τομέα αυτό. Μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε την προσοχή μας εξάλλου και στη λεγόμενη εδαφική ατζέντα την ε, αξιολόγηση αυτής της ατζέντα και των λεγόμενων εδαφικών προοπτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εδαφική ατζέντα και η εξέτασή της, η παρεξέτασή της είναι πάρα πολύ σημαντική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των προσπαθειών μας. Αυτή η ατζέντα η οποία ενεκρίθη το έτος 2007 δεν έχει εκπληρώσει τις προσδοκίες οι οποίες είχαν τότε δημιουργηθεί. Ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα λοιπόν της Ουγγρικής Προεδρίας θα πρέπει να είναι να υπάρξει μια περαιτέρω επανεξέταση και εξέλιξη της εδαφικής ατζέντα και στα πλαίσια αυτής της επανεξέτασης θέλουμε να θέσουμε έμφαση στην εδαφική σχεδίαση, την εποπτεία και τη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και την περαιτέρω εξέλιξη αυτής της πολιτικής. Στα πλαίσια αυτής της εδαφικής ατζέντα θέλω να επιστήσω την προσοχή σας και στο γεγονός ότι εάν θέλουμε να έχουμε μια εποφελή στρατηγική ε, Ευρώπης 2020 είναι πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν μέσα στο πλαίσιο αυτό. Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν λοιπόν όλα αυτά τα πολύπλακα εγχειρήματα χρειάζεται να υπάρξουν εξελίξεις σε πολλούς τομείς και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές από τα κράτη-μέλη. Είναι απαραίτητο η, η πολιτική συνοχής να παίξει κάποιο ρόλο και μέσα στα πλαίσια της επιζήτησης της εδαφικής συνοχής. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε ότι στα πλαίσια αυτής της πολιτικής και η επόμενη προεδρία, η πολιτική προεδρία, θα έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναπτύξουμε επιμέρους πολιτικές, να υπάρξει σχεδιασμός και οργάνωση της εφαρμογής των πολιτικών αυτών. Η αξιολόγηση των επιτευγμάτων της περιφερειακής πολιτικής επέχει επίσης ένα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η εδαφική ατσέντα θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σημαντικότερο εγχείρημα για μας είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να αναπτυχθούν ε, περαιτέρω προγράμματα τα οποία θα ισχύουν και μετά από το 2013. Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου μπορεί να υπάρξει θετική συνεργασία εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει και τις προτάσεις της σε σχέση με την ε, νομοθετική ρύθμιση τον Ιούνιο 2011 για την πολιτική συνοχή. Ε, και θα ήθελα να ζητήσω από τη δική μας πλευρά την υποστήριξή σας για το έργο της Ουγγρικής Προεδρίας. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προετοιμασία της επόμενης φάσης της πολιτικής συνοχής. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η αποτελεσματική σας υποστήριξη. Θα ήθελα εν κατακλείδη να σας πω ότι το μήνυμα και το σύνθημα της ε, Ουγγρικής Προεδρίας είναι ότι χωρίς μια συνοχή των περιφερειών και των κρατών της Ευρώπης δεν μπορεί να υπάρχει Ευρώπη και φυσικά χωρίς αυτήν την ε, συνεργασία δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνιστική και ισχυρή οικονομία. Χρειάζεται λοιπόν η συνοχή αυτή την ανταγωνιστικότητα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω να επικράτησε τόση σιωπή κατά διάρκεια συνεδριάσεων αυτή τη Επιτροπή. Μα δώσετε όμω ιδιαίτερη τροφή προ Και είμαι βεβαία πω οι συνάδελφοι θα έχουν πολλά σχόλια και ερωτήσει να σε υποβάλουν. Η συντονίστρια τη οριστική Ομάδα τώρα. Αν μπορώ να ξεκινήσω με την τελευταία σας φράση Είπατε ότι χωρίς πολιτική συνοχής, ισχυρή πολιτική συνοχής δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτή την περίπτωση γιατί το πρόγραμμα της ε, Ουγγρικής Προεδρίας το οποίο πήρα στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα δεν αναφέρει καθόλου τη λέξη συνοχή. Η λέξη πολιτική συνοχής δεν αναφέρεται ούτε άπαξ στο πρόγραμμα αυτό το μόνο το οποίο έχει κάποια σχέση με την πολιτική συνοχή είναι η αναφορά τη στρατηγική για το Δούναβι, την περιφέρεια του Δούναβι. Κατανοώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ουγγαρία, αλλά θα ήμουν πολύ πιο ευτυχισμένη αν υπήρχε εδώ στην κατάλληλη θέση η πολιτική συνοχή όπω το έχετε παρουσιάσει τώρα εξάλλου. Εγώ συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία μαζί σα απόλυτα. Αυτά που αναφέρατε ω αναγκαιότητε που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Μα Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή. Ερχόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Και γι' αυτό με ενδιέφερε πάρα πολύ τι θέλετε να κάνετε μέσα στο επόμενο εξάμεινο ώστε να διαμορφωθούν οι μελλοντικέ δημοσιονομικές προπτικές επέκεινα του 2013 και να προετοιμαστούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Ποιες προτάσεις έχετε για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Μιλήσατε ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ συνοχής και τομεακής πολιτικής. Σημαίνει για σας ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι μπορεί να υποστηρίξετε μια, ένα κατακαιρματισμό της πολιτικής συνοχής σε πολλούς επιμέρους τομείς ή θέλετε να έχετε μια ισχυρή πολιτική συνοχή η οποία θα, δεν θα κατακαιρματιστεί σε διάφορους τομείς. Και κάτι ακόμα το οποίο δυστυχώ δεν αναφέρεται. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αρχή αυτή τη εταιρικότητα, δηλαδή η συνεργασία τοπικών περιφερειακών αρχών και άλλων φορέων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μελλοντική διαμόρφωση της πολιτικής συνοχής. Και κάτι άλλο θα ήθελα να ακούσω από τα χείλη σας. Μίλησατε πάρα πολλές φορές για την απλοποίηση των διαδικασιών. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς επί χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, θα το λέμε πάρα πολλά χρόνια. Έχετε εσείς ως Ουγγρική Προεδρία κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις να μας παρουσιάσετε και ακόμα που μπορούσαν να υλοποιηθούν στην τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικού σχεδιασμού ή είναι απλώς μια πρόγευση για τις μελλοντικές δημοσιονομικές σχεδιάσεις. Ευχαριστώ, Ο Σουρίαν τώρα, παρακαλώ. Το ερώτημά μου σχετίζεται με το προηγούμενο. Στην Επιτροπή Προπολογισμού κάνουμε προσπάθειες προκειμένου να προωθήσουμε και την πολιτική συνοχή και να την υπερασπιστούμε. Και η χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση πολιτική συνοχή πολύ συχνά κατηγορούμεθα. Ναι, μα λένε, αλλά, αλλά το ελεκτικό συνέδριο διαπίστωσε πολλά λάθη, βρήκε πολλά λάθη αν θέλετε και πολλές αν θέλετε ατασταλίες στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Πολλά από τα λάθη αυτά κατά τη γνώμη μου πάντως οφείλονται αν θέλετε στη γραφειοκρατία, στο δαίμονα της γραφειοκρατίας και πολύ συχνά οι ετούντες, αυτοί που κουβάλλουν τι αιτήσει δηλαδή, είναι υποχρεωμένοι να θέλετε να συμπληρώσουν αν θέλετε γελίες ερωτήσεις Πολλές φορές αν θέλετε υπάρχουν και υπόνοιες περί διαφθοράς, περί δωροδοκίας, περί χρηματισμού κτλ. και πάει λέγοντα. Τι έχει κατά νου η Προεδρία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κριτικές και τις επικρίσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Γι' αυτό λοιπόν ε, η παρατήρηση συναδέλφου προηγουμένω περί απλοποίηση, δηλαδή ότι αυτό θα καταστήσει, αν θέλετε, και διαφανέστερο τον κανονισμό και αυτό θα κάνει πιο εύκολο το έργο μα στην Επιτροπή του Προπολογισμού και θα είναι μια πολύ πιο εύκολη αν θέλετε για μας να υπερασπιστούμε και να περαμηθούμε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Βλάσικ τώρα. Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μας, καταρχήν. Χαιρετίζω επίση και τη δυνατότητα που μα προσφέρετε να απευθύνω κάποιε ερωτήσει. Εκτιμώ το γεγονό ότι αναφερθήκατε στην σημασία τη ολοκλήρωση αυτών των υποδομών και τη συμπλήρωση αυτών των υποδομών που απαιτείται βεβαίω στα νέα κράτη-μέλη διότι αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη συνολικά. Στην αρχή όμω επίση αναφερθήκατε σε συγκεκριμένε πτυχέ αυτή τη πολιτική συνοχή. και αναφερθήκατε και στου στόχου. Μπορείτε θα μπορούσατε να τα περιγράψετε όλα αυτά με περισσότερε λεπτομέρειε. Δεύτερο ερώτημα. Αναφερθήκατε και αναφέρατε και πολύ καλά κάνατε στην σημασία της σχέση που πρέπει να υπάρχει με την ε, τοπική αυτοδιοίκηση, τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές σε ό,τι αφορά τη συζήτηση αν θέλετε, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη. Όταν είδα δηλαδή τις προτάσεις που κάνατε για τις σημαντικές εκδηλώσεις που προτίθεστε να οργανώσετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, δεν βρήκα πουθενά να υπάρχει τίποτα, να προβλέπετε και να οργανώσετε δηλαδή κάποια συνάντηση του είδους αυτού. Και προ όφελο αν θέλετε, αυτών των περιφερειακών αρχών. Ε, μια συνάντηση δηλαδή της Προεδρίας για αυτόν τον περιφερειακό αρχών, αν θέλετε, σε αυτό το φόρουμ δηλαδή που θα γίνει πριν τα τέλη Ιανουαρίου. Προβλέπετε να γίνει κάτι τέτοιο, έχετε κατά νου μια τέτοια πρόταση. Παρακαλώ. Απαντήσατε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Επόμενο μιλήτρια. Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Έχω πολλές ερωτήσεις. Χαίρομαι που η αστική αν θέλετε διάσταση αποκτά μεγαλύτερη σημασία και ελπίζω να την ξαναβρούμε στις εκδηλώσεις. Μια πραγματική αν θέλετε αστική ατζέντα της Ουγγρικής Προεδρίας θα θέλαμε να υπάρχει. Για πολλά πράγματα. Αφενός πρέπει σήμερα να αναρωτηθούμε το εξής η θέρμανση του πλανήτη και τι ρόλο θα δώσετε στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τι επιφυλάσσετε. Πώς αν θέλετε θα τονίσετε και θα επισημάνετε αυτή την προβληματική και αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, μιλήσατε για τη διακυβέρνηση σήμερα, ολονά και περισσότερο. Η Επίτροπος αν υπερασπίζεται το ρόλο των πόλεων, έχετε εσείς το ίδιο όρομα με αυτήν διότι θα απελευθερώσουν αν θέλετε το, τον πιλότο, οι πόλεις γιατί η καταπολέμηση αν θέλετε τις θέρμανση και η προσπάθεια που γίνεται για το κλίμα γίνεται μέσω των πόλεων. Θα προβλέπετε αν θέλετε νέα χρηματοδότηση, καινούργια χρηματοδότηση για τις πόλεις. Και να θέσω και ένα άλλο ερώτημα πολύ σοβαρό όσον αφορά του δείκτε. Προέρχομαι από μια περιοχή, αν θέλετε, ονομάζεται, που είναι μια από τι πλουσιότερε στην Ευρώπη. Και παρόλα αυτά οι ανισότητες εντός αυτής είναι ολοένα και αυξανόμενες. Επομένως το ερώτημά μου είναι σαφές και ξεκάθαρο. Σήμερα, τη σήμερα ημέρα δηλαδή, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, θα ξαναδείτε αυτή την έννοια, αν θέλετε, του καθαρίστου χωρίου προϊόντος, του ΑΕΠ, που για μένα δεν αποτελεί, αν θέλετε, ένα καλό ορισμό, αν θέλετε, για να χαρακτηρίζει τις περιοφέρειες αλλά έχετε αν θέλετε πρόθεση να ξανανοίξετε το θέμα αυτό, να βάλετε ένα νέο ορισμό στο τραπέζι και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο τον ε, κύριο Υπουργό να απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, Καλώ ήλθατε κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε τη Ουγγρική Προεδρία στην Επιτροπή μα. Αν και η επίσημη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μελλοντικό σχέδιο της πολιτικής συνοχής θα παρουσιαστεί τον πιο πιθανό επί Πολωνικής Προεδρίας, η χρονική περίοδος της Ουγγρικής Προεδρίας θα είναι πολύ καθοριστική για την εξαγωγή συζητήσεων στρατηγική σημασία αναφορικά με το μελλοντικό προσανατολισμό της πολιτικής συνοχής. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας θα αποτελέσει στρατηγικό συνομιλητή σε αυτές τις συζητήσεις. Κύριε Υπουργέ, έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς βλέπετε την πρόταση της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή για την εξάρτηση της αποταμίευσης των πόρων των διαφορετικών ταμείων από την τήρηση μακροοικονομικών προϋποθέσεων. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και θα το υπερασπιστείτε στα πλαίσια των στρατηγικών συζητήσεων. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πώς βλέπετε την μακροπεριφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Θα υποστηρίζετε για παράδειγμα την ανάγκη για διάθεση κονδυλίων ειδικά για τέτοιου είδους στρατηγικές ή πιστεύετε ότι το τρέχον πλαίσιο είναι επαρκές για την στήριξη αυτής της μορφής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Υπουργό, για τα ερωτήματά σα. Για να είμαι ειλικρινή μαζί σα, κυρία Κρέλ, αυτό το οποίο είπατε για την ε, απουσία της έννοιας συνοχής στο ουγγρικό πρόγραμμα Το μόνο το οποίο μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω αυτά που είπα εγώ στα εισαγωγικά μου σχόλια. Και με τη συνείδηση μου ήσυχη μπορώ να το πράξω αυτό. Στις 7 Νοεμβρίου όταν ε, συνάντησε η Ουγγρική κυβέρνηση την Κομισιόν και τον ε, Ιανουάριο που επαναλήφθηκε αυτή η συνάντηση και στις δύο ευκαιρίες η πολιτική συνοχή ήταν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε. Ακόμα έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι για την Ουγγρική Προεδρία είναι τόσο σημαντική η πολιτική συνοχή. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω, να το επαναλάβω και να το τονίσω και πάλι. Και για μας, το ξαναλέω, η πολιτική συνοχή είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία. Και υπάρχουν δύο βασικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένα είναι η παραδοσιακή ολοκλήρωση και η αλληλεγγύη και το δεύτερο, δεύτερος πυλώνας είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται την ενίσχυση και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της και στις δύο περιπτώσεις είναι σημαντικό εργαλείο η πολιτική συνοχή. Θα παραμείνει λοιπόν πάρα πολύ σημαντική μέσα στο πρόγραμμα της ουγγρικής πολιτικής και νομίζω ότι είναι μια πολιτική η πολιτική συνοχή η οποία θα πρέπει να διατρέχει οριζόντια όλα τα προγράμματα και όλες τις κατευθύνσεις. Και αυτό φυσικά, όπως είπα, συνδέεται και με τα ζητήματα της δημιουργίας υποδομών και επίσης το γεγονός ότι η πολιτική ε, συνοχής θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση να αντιμετωπίζεται όχι μονάχα στον τομέα αυτών της ε, εδαφικής συνοχής αλλά και της ανταγωνιστικότητας, της σύγκλησης με, σε υψηλούς βαθμούς ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό λοιπόν το τμήμα του προγραμματός μας, αυτό θέλω να σας πω, πιστέψτε με, η πολιτική συνοχής είναι μια σημαντική κατεύθυνση μέσα στο πρόγραμμα της ε, Ουγγρικής ε, Προεδρίας. Αυτό συμπεριλαμβάνεται και στη στρατηγική μας για τον Δούναβη, για τους Ρωμά. Έχουμε υπογραμμίσει αυτές τις προτεραιότητες μέσα στο πρόγραμμα της Προεδρίας. Επίσης, μπορώ να σας δώσω μια απάντηση σε σχέση με το σχεδιασμό για τα δημοσιονομικά στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. για μας για το θέμα της ε, κατατομής κατάτμισης της ε, περιφερειακής πολιτικής είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με, με τις υποδομές, με, την, ε, με τις ενεργειακές υποδομές και με άλλων μορφών ε, υποδομές επικοινωνιών κτλ. Όλα αυτά φυσικά έχουν σημαντικές ανάγκες. Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν με την πολιτική συνοχή. Εγώ θεωρώ ότι το περιθώριο το οποίο έχει στη διάθεσή της η Προεδρία στους επόμενους έξι μήνες σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές πέραν του 2013 είναι πρόφανως περιορισμένες μέχρι το 2013 τουλάχιστον περιορισμένε, εμεί θα πρέπει να λειτουργήσουμε μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του ΕΚΟΦΗΝ. Αυτό δεν έχει να κάνει με τι ε, επιμέρου πολιτικέ. Οι πολιτικέ αυτέ φυσικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε και το γενικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Η θέση της Ουγγρικής Προεδρίας είναι ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να διατηρήσουμε το ειδικό βάρος της πολιτικής συνοχής μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρήσουμε και την πολιτική της αξία. Ο προϋπολογισμός φυσικά είναι σημαντικός και γι' αυτό πρέπει να διατηρηθεί η συμμετοχή της πολιτικής συνοχής μέσα στον προϋπολογισμό προτεραιότητες μας λοιπόν θα είναι αυτές και σας λέω και πάλι ότι μετά από την Ουγγρική Προεδρία θα αναλυφθεί η σκητάλη και από την Πολωνική Προεδρία. Ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό έχω απαντήσει όχι ένα, αλλά πολλά ερωτήματα που μου τέθηκαν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στους πόρους της ε, πολιτικής συνοχής και σε σχέση με τους μηχανισμούς αυτής της πολιτικής. Τώρα, για το συγκεκριμένο σας ερώτημα, για τις αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν μετά από το 2014, θα πρέπει να γίνουν μετά από μια ενδελεχή εξέταση των διαφόρων συστημάτων και των διαφορετικών χρονικών περιόδων που θα ισχύουν αυτά τα συστήματα και το να προκαταλάβω αυτή τη διαδικασία μπορεί να είναι και βλαβερό πιστεύω στην πράξη. Αυτό λοιπόν ισχύει για το μέλλον, ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τη μακροχρόνια εξέλιξη της πολιτικής συνοχής πολύ προσεκτικά. Η ελπίδα μας είναι ότι οι άτυπες υπουργικέ σύνοδοι του Μαΐου η σύνοδος μάλλον του Μαΐου θα μπορέσει να μας βοηθήσει να καταλήξουμε και σε μια ευρύτερη συνένεση σε σχέση με την κατεύθυνση που πρέπει να λάβει η πολιτική συνοχή στο μέλλον. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα οποία εξαρτώνται από αυτό το ζήτημα και περιθωριακά θα ήθελα να σας πω ότι το θέμα της αιρεσιμότητος που συνδέεται με το θέμα αυτό γιατί η λογική όλου του συστήματος θα πρέπει να επανεξεταστεί θα πρέπει να μας οδηγήσει οι πόροι, στο, οι που θα είναι στη διάθεσή μας να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο αλλά στη συνέχεια να εφαρμοστούν και να κατευθυνθούν στους τομείς όπου είναι απαραίτητοι με την διατήρηση της διαφάνειας. Αυτά που είπε τώρα ο κύριος, σε αυτά που είπε ο κύριος Σούριαν για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Βάσει της έκθεσης του 2009, ο, το επίπεδο των σφαλμάτων έναντι του 2008 έχει μειωθεί τα μάλα. Αυτό δείχνει ότι το ισχύον σύστημα στη βάση του λειτουργεί πολύ καλά και έχει τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξη. Γι' αυτό η υπεποίθησή μου είναι ότι τα μέτρα τα οποία έχουν αναλυφθεί από την Κομισιόν σε σχέση με τον μελλοντικό προγραμματισμό μπορούν να μας δώσουν εμπιστοσύνη σε σχέση με το μέλλον του συστήματος. Το σύστημα φυσικά χρήζει περαιτέρω εξέλιξης χωρίς αυτό να οδηγήσει σε ριζικές ανατροπές. διότι το σύστημα ήδη ενέχει τις δυνατότητες βελτίωσης στο εσωτερικό του ήδη. Και οι βελτιώσεις αυτές θα πρέπει να, να τύχουν εκμετάλλευσης. Δεν είμαστε λοιπόν επαναστατικοί σε σχέση με τις αλλαγές που θεωρούμε ότι πρέπει να επιτευχθούν. Πιστεύω ότι και τώρα περνάω στο επόμενο ερώτημα το οποίο τέθηκε που είναι το θέμα του, της καταμέτρησης του ΑΕΠ όπως αναφέρθηκε εμείς υποστηρίζουμε αλλά τη χρήση του ΑΕΠ γνώμονος. Εμείς υποστηρίζουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την διατήρηση των ε, ισορροπιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η Ουγγρική Προεδρία δεν υποστηρίζει λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει το ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη θα θελήσουν ενδεχομένως να προτάξουν άλλους δείκτες και όχι απλώς το, το, το ΑΕΠ ως έχει σήμερα. Εμείς θέλουμε να έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σύστημα δικτών το οποίο να είναι συνολικό και να ισχύει για όλους, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη δυνατότητα σε εθνικό επίπεδο να χρησιμοποιείται ή και σε περιφερειακό ενδεχομένω επίπεδο να χρησιμοποιείται ένα άλλο σύνολο από δείκτες. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω στα σημεία αυτά. Και μπορούμε να διαπιστώσουμε επίσης ότι και το ζήτημα των, ε, της συνεργασίας με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, όπως τονίστηκε και από το βιβλίο Βλάσεκ, είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων και η ελπίδα μας είναι ότι θα τύχει πρέπουσα εξέταση στο θέμα αυτό στην άτυπη συνόδο του Μαΐου. Και θα έχω την κατάλληλη μέρημνα ώστε στην, στην ε, σύνοδο αυτή θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό ενδελεχώς. Σας υπόσχομαι ότι θα είναι στην ημερησία διάταξη το θέμα αυτό. Μόνο όταν αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα πλήρως θα μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ένα πλήρες πλέγμα μέτρων και συμφωνεί η Ουγγρική Προεδρία να υπάρξει στα πλαίσια της ε, πολιτικής συνοχής μία ε, αύξηση της εδαφικής ε, συνοχής και μέσα σε αυτό οι αστικοί χώροι παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Μας, μας είναι προφανές ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργηθεί το απαραίτητο πλαίσιο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά αυτές οι πόλεις. Η Ουγγρική Προεδρία θα συνεχίσει την πρωτοβουλία της Βελγικής και Ισπανικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά την εδαφική συνοχή για τις πόλεις, ότι οι πόλεις, δηλαδή οι αστικοί σχηματισμοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως περιφέρειες και επομένως θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την περαιτέρω εξέλιξή τους. και αυτή θα είναι και η αντιμετώπιση που θα ακολουθήσει η Ουγγρική Προεδρία. Επίσης, στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε και την πολιτική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. και ήμουν παρόν σε μια ακρόαση στην, ε, σε μια για την κλιματική αλλαγή και είχα παρουσιάσει πλήρω τι προτεραιότητε τη Ουγγρική Προεδρία για το θέμα τη αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων τη κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στι επερχόμενε δεκαετίε που πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από το οποίο θα προσδιοριστεί και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η πολιτική για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά κριτηρίων. Κάθε επιμέρους πολιτική θα πρέπει να έχει και την πτυχή της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει επομένως να ενσωματωθεί πλήρως και αυτή η πτυχή της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής στην πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ξέρετε όλοι ότι η πολιτική έναντι της κλιματικής αλλαγής είναι ένας χώρος στον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε επί πολλούς μήνες και ίσως έτη τις προσπάθειές μας μετά από την πρόσφατη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταλήξει σε μια ενιαία αντιμετώπιση η οποία μετά θα ενσωματωθεί στις πολιτικές της. Είναι λοιπόν μια πολιτική η οποία θα πρέπει να ξεσφα... μια σειρά αποφάσεων πρέπει να εξασφαλίσει την γεφύρωση των πολιτικών μας και είναι γεγονός ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χώρο ευρωπαϊκό, ο οποίος βασιζόμενος στην πολιτική συνοχή μπορεί να έχει ένα πιο ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Περαιτέρω νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και για την ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης εν γέννη. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν τις δυνατότητες που παρέχονται από την ε, περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις περιφέρειες μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός όπως ανέφερα προηγουμένως, όλα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν στην πολιτική ε, συνοχής. Είναι σημαντικά βήματα. Ένα περαιτέρω ερώτημα το οποίο ετέθη είναι το θέμα της εταιρικής σχέσης που πρέπει να εξασφαλίσουμε σε περιφερειακό και σε τοπικό επίσης επίπεδο. Να μπορέσει λοιπόν αυτή η εταιρική σχέση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους φορείς τους αντίστοιχους να ενσωματωθεί στην πλήρη πολιτική συνοχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ακόμα 15 λεπτά που μας έχουν απομείνει. Περάσουμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Παρακαλώ, εστε σύντομοι και θα έχει την ευκαιρία μετά ο Υπουργό να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ε, Καταρχάς να σας συγχαρώ για την προσέγγιση που είχατε πάνω στο ζήτημα της πολιτικής συνοχής ε, όπου και τονίζετε τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει στο μέλλον. Ε, το ερώτημά μου αφορά στην εδαφική συνοχή. Στο έγγραφο που λάβαμε αναφέρεστε στους ε, στόχους αλλά και τα διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη της Προεδρίας σας για την εδαφική συνοχή, μιλάτε για θέματα χωροταξίας, για την εδαφική ατζέντα κλπ. Συγκεκριμένα αυτά πράγματα μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με την άποψη της Ουγγρικής Προεδρίας αναφορικά με την εδαφική πτυχή στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ουγγρική Προεδρία δεν επιθυμεί να διαχωρίσει το θέμα του κοινωνικού ταμείου ε, την πολιτική συνοχή. Ε, έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση σε ό,τι αφορά την ε, διασυνοριακή πολιτική. Αναφερθήκατε σε πολλές πτυχές, αλλά δεν αναφερθήκατε σε αυτήν την ε, διασυνοριακή περιοχή. Υπάρχουν περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, συχνά πρόκειται για τις ε, φτωχότερες περιοχές. Εδώ πρέπει να βρούμε λύσεις συγκεκριμένες. Υπάρχουν κάποια μέτρα, κάποια εργαλεία μέσω των οποίων προτίθεται να στηρίξει η Ουγγρική Προεδρία αυτές τις ε, περιοχές. Δεύτερη ερώτηση, το θέμα της ανεπιβημένης προβολής ορατότητας, αν θέλετε, της πολιτικής συνοχής. Θα ήθελα να γνωρίσω ποιες είναι οι δράσεις ε, που η Ουγγρική Προεδρία προτίθεται να αναλάβει ώστε να υπάρξει καλύτερη προβολή της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αγκουράκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις να κάνω στον ε, κύριο Υπουργό. Η πρώτη είναι εξή. Έκανε λόγο στην εισήγησή του για την ανάγκη θέσπισης κάποιων κριτηρίων ώστε να φαίνεται η απόδοση της πολιτικής συνοχής. Χρειαζόμαστε δηλαδή κριτήρια για να δούμε εάν αποδίδει πολιτική συνοχής. Αν κατάλαβα καλά τη μετάφραση. Έχει κάτι υπόψη το κύριο Υπουργό τι, τι είδους κριτήρια θα μπορούσαν να ήταν αυτά. Και μια δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει ε, με, το, ε, με το θέμα των κυρώσεων. Είπε ο κύριο Υπουργό ότι στα θέματα των κυρώσεων για τα σφάλματα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Συμφωνώ απόλυτα. Επειδή και ο κύριο Σταυρακάκη έθωσε ένα ερώτημα και δεν ακούσαμε κάτι, Μήπω μπορεί να επανέλθει στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ κύριε κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η χώρα σας όπως και η δική μου, η Ελλάδα, είναι από αυτές που έχουν πληγεί σοβαρά από την ε, οικονομική και κοινωνική κρίση. Παράλληλα, η περιβαλλοντική κρίση συνεχίζεται, συνεχίζεται να επιδεινώνεται και δεν περιορίζεται στην κλιματική αλλαγή όπως γενικόλογα αναφέρατε πιο πριν. Η Κομισιόν εκτιμά σε κείμενό της με τον ίδιο τίτλο ότι η περιφερειακή πολιτική συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη του 2020. Αναφέρει μάλιστα συγκεκριμένα ότι υπάρχουν τρεις προτεραιότητες. Μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοπικιλότητας, οικολογική καινοτομία. Αυτό σημαίνει πράσινες επενδύσεις και νέες πράσινες θέσεις εργασίας, που οι πράσινοι τις υπολογίζουμε σε 5 εκατομμύρια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς, ως Ουγγρική Προεδρία, ποιες προτεραιότητες σχεδιάζετε να προωθήσετε στην περιφερειακή πολιτική σε αυτούς τους τομείς, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσει για πολιτικές που να συνδυάζουν ταυτόχρονη διέξοδο τόσο για την οικονομία όσο και για το περιβάλλον. Thank you, Thomas Deutsch. Eh, eh, Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ στην Περιφερειακή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνώρισα τον κύριο Υπουργό πριν από 24 χρόνια και τότε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε όταν η Ουγγαρία ήταν ακόμα στο κομμουνιστικό στρατόπεδο δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι σήμερα θα εμφανιζόσασταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Ουγγαρία σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν τότε αδιανόητο κάτι τέτοιο. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άποψη αυτή νομίζω ότι είσαστε πραγματικά το κατάλληλο άτομο για να συζητήσει αυτά τα θέματα κύριε Υπουργέ. Το πρόγραμμα το οποίο έχετε παρουσιάσει το χαιρετίζω, εγώ συμφωνώ με το γεγονός ότι ο στόχος της μάλλον, η στόχη της Ευρώπης 2020 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν προγράμματα μεταρρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης οι διάφορες περιφέρειες πρέπει να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι περιφέρειες θα παίξουν ένα πιο σημαντικό ρόλο μέσα στη διαμόρφωση πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το να σας συγχαρώ για την θαυμάσια παρουσίασή σας και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Ουγγρική Προεδρία. Όπως ξέρετε, στο χρονικό διάστημα 2007-2013 η περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κονδύλιο του ε, προϋπολογισμού με συνολική χρηματοδότηση για τα 7 χρόνια 380 δισεκατομμύρια. Αυτό δείχνει και τη σημασία του είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να καταμαρτυρήσω ο ίδιος γιατί έρχομαι από μια μικρή ε, νησιωτική περιφέρεια την Μαδέρα στην Πορτογαλία που πριν από 30 χρόνια βρισκόταν σε ΑΕΠ 40% περίπου του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη στις βοήθειες που πήρε ιδίως από το Ταμείο Συνοχής κατάφερε να μειώσει την απόστασή της από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 96% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ΑΕΠ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός καλού μαθητή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρέμβασή σας κύριε Υπουργέ αναφερθήκατε ιδιαίτερα στο θέμα της διακυβέρνησης. Θέλω να σας θέσω ένα απλό και άμεσο ερώτημα. Με ποιο τρόπο η Ουγγρική Προεδρία θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής με το να έχει μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, να έχει πιο ευέλικτα προγράμματα και να προωθήσει τις πρωτοβουλίες που γίνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κύριε Σενέμ, ευχαριστώ δηλαδή. Κυρία Σρέντα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, και εγώ θέλω να κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο ερώτημα και να αναφερθώ σε ένα μικρό θέμα που αναφέρατε στο πρόγραμμά σας η στρατηγική του ε, Δούναβη είναι ένα από τα αγαπημένα σας παιδιά και είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για όλους μας από δύο πτυχές. Καταρχήν, γιατί κατάλαβα ότι είναι σημαντικό το θέμα του περιβάλλοντος και το θέμα της πλοημότητος του Δούναβη παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Στα πλαίσια αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά και επίση υπάρχουν και νέα στοιχεία τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη στρατηγική του Δούναβη, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία σε επίπεδο ε, μακροπεριφέρειας και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Το ερώτημά μου είναι πού θα βρείτε τη χρηματοδότηση για αυτό το πρόγραμμα. Έχετε σκέψεις για το να γίνει κάποια αναδιανομή των κονδυλίων μεταξύ των περιοχών του στόχου 1 του στόχου 2 και του στόχου 3. Λέτε θέλουμε να έχουμε περισσότερο χρήμα για το στόχο 3 επειδή έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά επιχειρήματα, εγχειρήματα. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχετε κάποιες ιδέες για την ανακατονομή κονδυλίων μεταξύ των διαφόρων στόχων. Ευχαριστώ. And the last question. Ο κύριος Όλμπρεχτ. Ελπίζω να είναι σύντομη η ερώτησή του. Πρώτα απ' όλα ω ευρωβουλευτή καταγόμενος από την Πολωνία να ευχηθώ ότι το καλύτερο στην Ουγγρική Προεδρία. Γιατί για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό η Προεδρία σας να είναι επιτυχής. Θα έχουμε μια ολόκληρη χρονιά δηλαδή χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μια ερώτηση τεχνικής φύσεως. Να ρωτήσω καταρχήν τον Υπουργό θα ήθελα το εξής. Θα ήθελα ο Υπουργό δηλαδή να μου πει ποια είναι η θέση τη Ουγγρική Προεδρία σε ό,τι αφορά το πόσα χρόνια θα πρέπει να διαρκούν αυτέ οι ευρωοπτικέ. 5, 7 ή 10 χρόνια, γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πολιτική συνοχή. Ξέρω βεβαίω ότι θα υπάρξουν διαπραγματεύσει. Θα ήθελα πάντω να γνωρίζω αν υπάρχει ήδη από τώρα θέση τη Ουγγρική Προεδρία. Ένα άλλο ερώτημα τώρα και πάλι τεχνική φύσεω να θέσω, αν μου επιτρέπετε. Θα θέλαμε να δούμε το πρώτο σχέδιο κανονισμών που αφορούν στην πολιτική συνοχή κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα, τη Ουγγρική Προεδρία δηλαδή, εννοώ. Ή θα θέλατε όλα αυτά να εμφανιστούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, αυτή τη στιγμή θα έχουν ληφθεί δηλαδή οι οικονομικέ ή δημοσιονομικέ αποφάσει. Γιατί την επόμενη Δευτέρα στο Φόρουμ για τη Συνοχή θα έχω μια συνάντηση και θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η προτίμηση τη Ουγγρική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προτού να απαντήσω στις ερωτήσεις, να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, αλλά και για τον ε, τρόπο με τον οποίο ε, δεχτήκατε τα σχόλιά μου και την παρουσίασή μου. Είμαστε, όπως ξέρετε, νέο κράτος και για πρώτη φορά αναλαμβάνουμε την Προεδρία. Αλλά θα δείξουμε, ελπίζω, πνεύμα ανοιχτό και ελπίζω να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση των προσδοκιών μας. θα απαντήσω σε όλους σας γραπτός, σε όσους, δηλαδή δεν έχω προλάβει να απαντήσω απόψε. Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι θα είμαι στη διάθεσή σας. Όποτε θελήσετε μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου Ξέρω ότι πολλά από όσα είπα χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση, αλλά δυστυχώ είχα μόνο ένα χρόνο, στο, ένα, μία ώρα συγγνώμη, στην διάθεσή μου και τα θέματα που μας απασχολούσαν είναι πολύ σημαντικά. Του των λεχθέντων θα ήθελα τώρα να προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που μου ετέθησαν. Πιστεύουμε πως ε, οι προϋποθέσεις και οι όροι παίζουν πολύ μεγάλη σημασία στην φορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Αυτό εξάλλου το ανέφερα και στην παρουσίασή μου, αλλά επιθυμώ να το τονίσω για μια ακόμη φορά και να ευεβεβαιώσω πως η ισότιμη μεταχείριση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο Η συμμεταχείριση λοιπόν θα πρέπει να υποστηριχθεί και να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να αλλάξει κανείς εν μέσω του ποταμού τις ε, βασικές συνθήκες και το πλαίσιο. Πρέπει να διατηρήσουμε τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουν κέρια σημασία μέσα στην κοινωνική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Αυτό ισχύει και για το σύστημα κυρώσεων. Δεν είναι θέμα του να αλλάξουμε το σύστημα, απλώς πρέπει να έχουμε τις προϋποθέσεις οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις διαδικασίες που έχουν στον τομέα αυτό. Πρέπει να είμαστε λοιπόν αυστηροί και Εγώ φυσικά ως πρόεδρος του Συμβουλίου δεν μπορώ να παρουσιάσω μονάχα την Ουγγρική θέση. Πρέπει να παρουσιάσω τη συνολική στάση του Συμβουλίου. Πρέπει να διαχωρίσουμε λοιπόν την προσωπική μου στάση, μάλλον την Ουγγρική εθνική θέση και την θέση του Συμβουλίου. Ο στόχος μας στο Συμβουλίο είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση η οποία θα οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων. Αυτό αφορά όχι μόνο και τις προϋποθέσεις, αλλά και τις βασικές θέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν και αυτό επομένως περιλαμβάνει και το ζήτημα της αιρεσιμότητας που είπατε προηγουμένως. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και να γίνει κατανοητό από όλους ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο βρίσκεται σε αρμονία με αυτά τα οποία θα αποφασιστούν σε επίπεδο δημοσιονομικών προοπτικών στο επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουμε και να έχουμε ένα κατάλληλο μηχανισμό διαχείρισης των κινδύνων, αλλά επίσης και για την ανάπτυξη περαιτέρω συστημάτων διακυβέρνησης που θα πρέπει να εφαρμοστούν στον τομέα της ε, συνοχής. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω απόλυτα το να υπάρξει μια σαφής διατύπωση της πολιτικής διακυβέρνησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να συνδέει την πολιτική συνοχής με το γενικό σύστημα, το γενικό δημοσιονομικό σύστημα. Εμείς έχουμε τονίσει την ανάγκη να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εργαστούμε προς τις κατευθύνσεις αυτές και η πολιτική συνοχής και η πολιτική εδαφική ατζέντα να ενισχυθούν και να ε, τροποποιηθούν, τροποποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετήσουν τους στόχους αυτούς. θέλουμε να δημιουργήσουμε και αυτές τις πράσινες θέσεις εργασίας. Και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και το έχουμε τονίσει και στο παρελθόν. Πρέπει σε όλες τις πολιτικές και στην πολιτική συνοχή συγκεκριμένα να εξασφαλίσουμε την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και είμαστε από αυτή την άποψη εξαρτώμενη από την αντιμετώπιση και της οικονομικής ε, κρίσης. Η οικονομική κρίση έχει μειώσει τις παραγωγικές δυνατότητες. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την αύξηση της απασχόλησης και την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τις παραγωγικές δυνατότητες που έχουν και αυτό μπορεί να γίνει και με την παροχή κινήτρων για ανάπτυξη περαιτέρω ανταγωνιστικότητας. Δεν είναι ο μόνος δρόμος, αλλά είναι ένας από τους δρόμους που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να βγούμε από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οικονομική κρίση. Εάν θέλετε να αναφερθείτε μπορεί να θέλετε να αναφερθείτε στους ανταγωνιστές μας στην Κίνα, στη Βραζιλία, την Ινδία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν κάτι κοινό στο επίπεδο της συνοχής και πρέπει και η Ευρώπη να εξασφαλίσει τη δική της πολιτική συνοχής. Και όπως είπα προηγουμένως η ορατότητα αλλά και η διαφάνεια θα ευνοήσουν την λειτουργία της ε, πολιτικής συνοχής. Και η απλοποίηση των διαδικασιών και η αναδιάταξη των προγραμμάτων είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για τη βελτίωση της ε, διαφάνειας στα εθνικά μας προγράμματα στο εθνικό μας πρόγραμμα μάλλον η Ουγγαρία το τελευταίο χρόνο έχει επιφέρει αλλαγές οι οποίες οδήγησαν στην ε, ενίσχυση της ε, διαφάνειας στη δική μας πολιτική, κάτι το οποίο ήταν θετικό για τη σύνολη πολιτική. Θελήσαμε λοιπόν να υπάρχει και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο σαφήνεια για το γεγονός ότι η πολιτική συνοχή είναι μια συνολική πολιτική, είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που μπορεί ο καθένας μέσα στο δικό του τοπικό χώρο να την πραγματοποιήσει. Είναι σημαντικό επομένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα νέα κράτη-μέλη, να μπορέσει να γίνει αντιληπτή να αντιληφτεί ως ένας θετικός φορέας πρόοδου. Για τη στρατηγική του Δούναβη τώρα. Θέλω και εδώ να πω κάτι ακόμα για το θέμα αυτό. Η άποψή μου είναι υπάρχουν τρία σοβαρά προγράμματα τα οποία τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Μάιο θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν σε συζητήσεις άτυπες μεταξύ Υπουργών όπου θα γίνει η κατάλληλη στόχοθεσία επί, των, επί τη βάση των προτάσεων της Ουγγρικής Προεδρίας και θα είναι ουσιαστικά μονογραφικές αυτές οι συναντήσεις μας για τα θέματα αυτά ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον τομέα της εδαφικής ατζέντα και, των, και της σωστής ερμηνείας της. Θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των Υπουργών για το θέμα αυτό. Δεν θέλω να προκαταλάβω το αποτέλεσμα το οποίο θα προέλθει. Ε, δεν ξέρω ποιες είναι οι απόψεις οι οποίες θα πρετανεύσουν, αλλά το Μάιο στην Υπουργική αυτή Σύνοδο και πριν από αυτήν την Σύνοδο θα, όταν θα έχει γίνει ήδη η συνάντηση των εμπειρογνώμων θα είμαι στη διάθεσή σας να επανέλθω και να λάβω το λόγο ενώπιόν σας για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και επίσης αυτό μπορεί να γίνει και μετά από την σύνοδο αυτή την άτυπη του Μαΐου. Και τέλος για τη στρατηγική του Δουνάβεως, θέλω να τονίσω ότι αυτή η στρατηγική για την Ογκρική Προεδρία δεν είναι μοναχα μία στρατηγική που στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά είναι και μία πολιτική που έχει να κάνει με τη μακροπεριφερειακή διάσταση της περιοχής συνάπτεται με την οικονομική ανάπτυξη και εάν δω την οπτική γωνία της δικής μου χώρας της Ουγγαρίας, φυσικά είναι πολύ σημαντική αυτή η πολιτική και για την ανάπτυξη του τουρισμού. Μας ενδιαφέρει η οικονομική πτυχή, η πλοημότητα δηλαδή του Δούναβη. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. η διαδικασία για την έγκριση της στρατηγικής του Δούναβη ξεκίνησε ήδη στις 19 Ιανουαρίου όταν έλαβε χώρα μια συνάντηση της ομάδας εργασίας για το θέμα αυτό. Η ελπίδα μας είναι ότι τον Ιούνιο αυτού του χρόνου στην ε, Σύνοδο του Συμβουλίου Κορυφής θα έχει περατωθεί η διαδικασία έγκρισης της στρατηγικής για το Δούναβη. Και ελπίζουμε ότι στο τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας θα έχουμε καταφέρει να κλείσουμε πλήρως το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν τα οποία είναι μακροπεριφερειακού χαρακτήρα πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα ενισχύσουν τη γνώση μας για τα θέματα αυτά ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε στο Συμβουλίο Κορυφής του Ιουνίου. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι εξ ονόματος όλων θα πρέπει να πω ότι εκτιμούμε και ευχαριστούμε για τις πολύ, αν θέλετε, καλές απαντήσεις που δώσατε στα ερωτήματά σας. Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας, είπατε ότι είστε δεθειμένος να είστε εδώ να μας ενημερώνετε, αλλά εξ ονόματος όλων των συναδέλφων να πω θα ήθελα ότι λογαριάζουμε στις προσπάθειες που καταβάλλετε, προκειμένου να εξασφαλίσετε, αν θέλετε, την σωστή, αν θέλετε, εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις εργασίες του Συμβουλίου γιατί εργαζόμαστε υπό το πρίσμα της νέας συνθήκης πλέον. Και αυτό νομίζω ότι ανοίγει, αν θέλετε, νέους δρόμους συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι αντιμετωπίζουμε πολλές και σημαντικές προκλήσεις που ενδιαφέρουν ε, τόσο εσά ως Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και εμά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν και για μια ακόμη φορά σα ευχαριστώ. Ευχόμαστε το καλύτερο και σα ευχόμαστε και δύναμη. Γιατί δεν θα είναι εύκολο πράγμα για εσά αλλά βεβαίω να ξέρετε ότι θα σας στηρίξουμε και στηρίζουμε τις προσπάθειε σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει και ο Ούγγρος Υπουργό. Before you go, I just have to announce that... Πρωτού φύγετε, πρωτού φύγετε. Το σημείο 6, η γνωμοδότηση Καρόνα δηλαδή, θα δούμε αυτό το ζήτημα μετά την ψηφοφορία αύριο. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν για το ζήτημα αυτό, αύριο μετά την ψηφοφορία